time. Right, if, if we could sit down, um... Συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσουμε για να μην χάσουμε πάρα πολύ χρόνο. He lost 10 minutes Ήδη έχουμε καθυστερήσει 10 λεπτά. Θα εξετάσουμε τα σημεία 6 και 7 της ημερήσιας διάταξης. Δηλαδή, δημόσια ακρόαση για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και επιχειρηματικού κεφαλαίου. Ο στόχος της ακρόασης αυτής είναι να μας βοηθήσει στην αξιολόγηση που θα κάνουμε. Δηλαδή είναι κατάλληλο το πλαίσιο που προτείνει η Επιτροπή για να υποστηρίξει τα ευρωπαϊκά αυτά ταμεία και τον τρόπο συλλογής κεφαλαίων το κάνει πιο αποδοτικό. ώστε να μπορέσει να βοηθήσει την, πρόταση, την πρόσβαση κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτά τα ίδια κεφάλαια και ως τύπου Έχουμε δύο μέρη. Θα χωρίσουμε πρώτα απ' όλα το πρώτο μέρος της ακρόασης στα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με εισηγήτρια την Σοφία Οκονή. Και έχουμε παρουσίαση του σχεδίου έκθεσής της, τις ε, δύο ομιλίες και για μία ώρα περίπου θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Η Σοφή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Σένινγκ, κύριο Ντόναχιου, χαίρομαι διότι θα σας μιλήσω σήμερα για αυτό το θέμα που εξετάζουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά και κυρίως για πρώτη φορά στα πλαίσια των ε, θεσμικών οργάνων που είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις και να δούμε πώς θα μπορέσουμε πριν να κάνουμε την ακρόαση για το ίδιο θέμα να δούμε τις βάσεις του θέματος αυτούς. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εξαιρετική. Είναι πάρα πολύ φιλόδοξη, το κείμενο είναι πολύ καλό και είναι και ένα διάβημα, αν θέλετε, το οποίο γίνεται πριν να... Euh, γίνεται πριν να αρχίσει η όλη διαδικασία. Δηλαδή να μπορέσουν να γίνουν προτάσεις εκ των προτέρων ώστε να μπορέσουν να, γίνουν, να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο ως διάβημα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ξέρουμε ότι για τις κοινωνικές επιχειρήσεις χρειαζόμαστε χρηματοδότηση των σύνων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι η κοινωνική επιχείρηση? Ο κύριος στόχος κοινωνικής επιχείρησης δεν είναι το κέρδος. Αυτό είναι σε δεύτερη θέση. Ο κύριος στόχος τους είναι να δημιουργήσει ένα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, δηλαδή εργατικές κατοικίες, ένταξη ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ατόμων στην κοινωνία, να βοηθήσει άτομα με κάποια αναπηρία, ένταξη των ε, αναλφαβήτων σε διάφορα προγράμματα. Για να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Φερρυπίν. Υπάρχουν κοινωνικά κομμωτήρια με franchise, δηλαδή έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κομμωτήρια άτομα τα οποία δεν έχουν αρκετά χρήματα, δεδομένου ότι σήμερα το κομμωτήριο κοστίζει ακριβά. Αυτά λοιπόν τα άτομα μπορούν να πάνε σε αυτά τα κοινωνικά κομμωτήρια που θα τα βοηθήσει να έχουν προς τα έξω όταν πάνε να ζητήσουν δουλειά μία καλή εικόνα. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο σήμερα αφορά το 10% των ευρωπαϊκών ε, επιχειρήσεων και περίπου 11 εκατομμύρια εργαζόμενους. Ποιος είναι ο στόχος της πρότασης κανονισμού? Ο πρώτος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σήμα, ένα διαβατήριο ευρωπαϊκό. για αυτά τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αυτά τα σήματα, τα διαβατήρια, θα είναι στη διάθεση των επενδυτών, των επαγγελματιών που θέλουν να κάνουν σε αυτό τον τομέα κάποιες επενδύσεις και να αναπτύξουν δραστηριότητες. Θα πρέπει επίσης ε, στον κανονισμό αυτό να πούμε ότι υπάρχουν κριτήρια τα οποία θα πρέπει να τηρήσει κανείς και αντιστοιχούν στις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων που σήμερα σχεδόν αποκλειστικά εξαρτώνται από επιχορηγήσεις και οι επιχορηγήσεις ξέρουμε ότι για να διονυστούν οι δραστηριότητες τέτοιων επιχειρήσεων δεν είναι πάντα σίγουρες και για να μπορέσουμε να τις εξασφαλίσουμε στον χρόνο θέλουμε να έχουμε έχουν αυτές τις επιχειρήσεις πρόσβαση και σε άλλες πηγές χρηματοδότησης. Τελείσαμε αυτό το ταμείο να είναι, εύκολα προσβάσιμο και ελκυστικό για τους επενδυτές, αλλά να προσφέρουν και μία κάποια ασφάλεια. Δηλαδή, η ευελιξία πρόσβασης να μην γίνει εις βάρος της ασφάλειας. Πρώτα απ' όλα, ελκυστικότητα, όπως σας είπα. Πιστεύουμε ότι το μέσον αυτό θα ήταν χρήσιμο εάν ήταν προσβάσιμα, εύκολο και ελκυστικό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κάτι το ευέλικτο, ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό επενδυτικών σχημάτων, το 70% του συνόλου της επένδυσης να αφορά αυτή την αλληλέγγυη επένδυση αν θέλετε. Καλό είναι αυτό το όριο, το κατόφλι. 100% θα ήταν ε, ε, ένα πολύ υψηλό ποσοστό, αλλά το 70% μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλό ποσοστό, πολύ καλό κατόφλι. Δεύτερο θέμα. Το θέμα της κοινοποίησης. Αυτό το μέσον δεν μπορεί να ισχύει παρά μόνο εάν ε, είναι δημόσια γνωστό και οι πάντες είναι ενημερωμένοι. Θα πρέπει λοιπόν οι, τα ταμεία αυτά να κάνουν την κατάλληλη ενημέρωση. Θα πρέπει να δούμε πολλές φορές αν μπορούμε για αυτό το θέμα να εμπνευστούμε από κάποια κράτη-μέλη, διότι ήδη υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία έχουν μια κάποια εμπειρία και πραγματογνωμοσύνη την κοινωνικέ επιχειρήσεις και θα ήθελα να υποφεληθούμε όλοι από την εμπειρία τους και τις θετικές τους εμπειρίες να τις συμπεριλάβουμε σε αυτό τον κανονισμό. Τώρα, η ασφάλεια. Ε, είπαμε ότι δεν θα πρέπει η πρόσβαση να γίνει εις βάρος της παροχής ασφάλειας. Εγώ θέλω να έχουμε διαφάνεια. Ο υπεύθυνο και διαχειριστής των ταμείων δεν θα πρέπει απλώς να είναι καταχωρημένος, αλλά θα πρέπει να πληρεί και τις προϋποθέσεις που χρειάζεται. Θα πρέπει επίση να ορίζουμε έναν θεματοφύλακα για κάθε είδους τέτοιου ταμείου με ευελιξία όπως είχε γίνει και για το IFM τις αγορές των χρηματοπιστωτικών μέτρων και να υπάρχει και η ε, νομική ε, προστασία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του κανονισμού, αυτό είναι το πρώτο στάδιο, θα πρέπει βραχυπρόθεσμα η Επιτροπή να μελετήσει και πολλά άλλα μέτρα και στην επόμενη εξέταση θα κάνουμε αξιολόγηση όλων αυτών των στοιχείων και θα δούμε κατά πόσον το κείμενο αυτό μπορεί να επεκταθεί. Θα πρέπει επίσης να δούμε ποιες θα είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις από την ύπαρξη και την δραστηριοποίηση αυτών των επιχειρήσεων, κάτι το οποίο μου φαίνεται ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και να δούμε μετά από την θέση σε ισχύ αυτού του κανονισμού όλα τα θέματα τα οποία θα πρέπει μαζί, βάσει της εμπειρίας, να αλλάξουμε, να ενημερώσουμε, ώστε να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση αυτού του ταμείου και χάρη, στον, των επενδυτών και υπέρ των επιχειρήσεων που θα είναι οι αποδέκτες αυτών των κονδυλίων. Ελπίζω ότι ήταν σύντομη και σαφής η παρουσίασή μου. Να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές που έκαναν πάρα πολύ θετική δουλειά κατά τη διάρκεια όλων των συζητήσεων, καθώς και τον Φιλίπ Λομπέρ, ο οποίος ε, έκανε την έκθεση για τα κεφάλαια κινδύνου, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια συνεκτική άποψη μεταξύ των δύο αυτών εκθέσεων που αφορούν κανονισμό και είμαι στην διάθεσή σας για να συζητήσουμε την έκθεση αυτή και με μεγάλη ευχαρίστηση θα ακούσω και τους εμπειρογνώμονες για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τώρα λόγο στους δύο μιλητές μας. Έχω πρώτα τον Νίκο Ντονόχιου CEO της Big Society Capital και τη Miriam Schoening. Ε, ε, Αν μπορείτε παρακαλώ να διατηρήσετε τα σχόλιά σας στα 5 λεπτά επειδή δεν έχω πολύ χρόνο και στη συνέχεια σας προειδοποιώ θα στραφώ στα μέλη για ερωτήσεις ε, στους σκιώδεις εισηγητής. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα έχουμε για τους σκιώδεις. Προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα πολύ γρήγορα, να εξετάσουμε τις εκθέσεις, τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Νίκ, έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω σήμερα. Σήμερα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω την Big Society Capital που είναι, βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο ως πρώτη τράπεζα με κοινωνικούς σκοπούς. Χρησιμοποιεί τους ε, ζήτητους τραπεζικούς λογαριασμούς για τη δημιουργία ενός κοινωνικού κεφαλαίου. Έχει μεγάλους ε, ε, εταίρους στην RBC, Barclays, Lloyds και SPC. Αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των κοινωνικών επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, με επένδυση σε ενδιάμεσους οργανισμούς κοινωνικών επενδύσεων. Αυτοί είναι οργανισμοί που διευκολύνουν και διοργανώνουν τη μεταφορά δανείων και άλλων επενδύσεων σε ε, οργανισμούς του κοινωνικού τομέα. Ε, οργανισμός κοινωνικού τομέα υπάρχει εξ ολοκλήρου ημερικός ε, προς όφελος της κοινωνίας αντί για την δημιουργία κέρδους για τους κατόχους και τους μετόχους του. Περιλαμβάνει φιλανθρώπικους οργανισμούς, κοινωνικές επιχειρήσεις, και διάφορες μορφές συνεργατικών, συνεταιριστικών επιχειρήσεων υπό ορισμένε συνθήκες. Μπορεί να, περιέχει, να περιλαμβάνει και εταιρείες κερδοφόρες. Επίσης, η DC θα κάνει μόνο επενδύσεις, όχι χορηγίες ούτε δωρεές. Για εμάς οι επενδύσεις μας θα πρέπει πάντοτε να δημιουργούν κάποια κοινωνική αξία θα χρειάζεται να επιτυγχάνουμε αποδόσεις τέτοιες ώστε να διασφαλίζεται η αηφορία της BSE και η μη εξάντληση του αρχικού της κεφαλαίου. Μου ζητήθηκε λοιπόν να περιγράψω τον τρόπο ανάπτυξη τη κοινωνική επένδυση στην Ευρώπη. Το να δημιουργήσουμε μια τέτοια αγορά χρειάζονται τρία πράγματα. Παροχή κεφαλαίου, ζήτηση για αυτό το κεφάλαιο και ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων που μπορεί να φέρουν μαζί την ε, παροχή, την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτή η κοινωνική αγορά για την οποία μιλάμε είναι ακριβώ έτσι. Θα σας μιλήσω λοιπόν για το καθένα από αυτά τα στοιχεία. Η παροχή κεφαλαίου σημαίνει ομάδες επενδυτών που επιθυμούν να κάνουν επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο. Πιστεύουμε ότι σήμερα υπάρχει βούληση για τέτοια επένδυση ωστόσο δεν έχει αξιοποιηθεί. Σύμφωνα με μια έρευνα στο Ηνωμένο Βασιλείο 65% θα ε, εξέταζαν το ενδεχόμενο μια τέτοια επένδυση, ωστόσο κανεί δεν την πραγματοποιεί. Ο, περισ... ο κυριότερο λόγο είναι ότι δεν γνωρίζουν πώ είναι αυτέ οι επενδύσει, πώ ορίζονται οι κοινωνικέ επιπτώσει ε, και τι απόδοση θα είχαν από μια τέτοια επένδυση. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν ε, αντιμετωπίζεται από ειδικού στις κοινωνικές επενδύσεις. Ε, συνεπώς επικροτούμε την πρόταση της Κομισιόν ε, για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Επίσης η Κομισιόν θα πρέπει να φροντίσει, να μεριμνήσει ώστε όλοι αυτοί να μπορούν να επενδύσουν σε αυτούς τους τομείς ανεξαρτήτως μεγέθους. Ε, καθώς αυτές οι επιχειρήσεις θα αυξάνονται ε, δεν γίνονται πιο εμπορικές. Συνεπώς, το να παρέχουμε κονδύλια μόνο σε μικρές επιχειρήσεις δεν βοηθούμε ε, την επιτυχία αυτών των επιχειρήσεων. Επίσης, ε, θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία επένδυση σε διάφορα μέσα, όπως τα νέα και τα καινοτόμα χρεόγραφα για την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων. Αυτά θα υποστηρίζονται επίσης ε, από εξαιρεσει που ε, βοηθούν σε πιο φθηνέ επενδύσει ε, σε καθοδήγηση από ρυθμιστικέ αρχές και ενδεχομένως φοροαπαλλαγέ σε τομείς όπου η απόδοση είναι χαμηλότερη από τη μέση της αγοράς. Αυτή η, αίτηση, η ζήτηση επένδυσης απαιτεί μια νομική δομή η οποία δεν υπάρχει απαραίτητα. Οι περισσότερε κοινωνικές επιχειρήσεις σήμερα εστιάζονται σε κοινωνικά αποτελέσματα. Ζητάει πρόεδρο από τον ομιλητή να μιλάει λίγο πιο αργά. Οι περισσότερε κοινωνικές επιχειρήσεις εστιάζονται στην παροχή κοινωνικών αποτελεσμάτων και όχι κερδών και σίγουρα όχι στη δημιουργία ασμάτων, ώστε να ε, δημιουργούν κέρδη οι μετοχοί τους. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις λοιπόν απαιτούν διαφόρους τύπους κεφαλαϊκής υποστήριξης. Απαιτούν ε, δανεισμό σε χαμηλά, με χαμηλά επιτόκια, αλλά απαιτούν επίσης και ε, κεφαλαιοποίηση μεσομετοχών. Συνήθως είναι ε, οι πιο δύσκολες μορφές ε, επένδυσης αυτές. Τέλος, ακόμη και αν υπάρχει προσφορά και ζήτηση και παρότι οι επενδυτές κατανοούν την κοινωνική επένδυση και οι κοινωνικοί οργανισμοί διαθέτουν τα μέσα για να λάβουν επενδύσεις, δεν θα υπάρξει αγορά εάν δεν υπάρχουν κάποιοι φορεί οι οποίοι θα συνδέουν όλους τους παρόχους ε, κοινωνικών κεφαλαίων, αυτοί που ονομάζουμε ενδιάμεση. Αυτό το ρόλο επιτελεί η BSC, η οποία παρέχει χρηματοδότηση, χρηματοδότηση για νέα ε, ταμεία κοινωνικών επενδύσεων, δημιουργεί νέες ε, καινοτόμες δομές συνεργασίας, όπως ομόλογα κοινωνικού αντικτύπου και οι κοινωνικές επιχειρήσεις ε, που επιθυμούν να ε, έχουν πιο αποτελεσματικές δραστηριότητες. Πρέπει να τονίσω και πάλι ότι πιστεύουμε ότι οι αγορές κοινωνικών επενδύσεων βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, δεν αντιμετωπίζουν όλα τα κοινωνικά προβλήματα που έχουμε, ωστόσο έχουν τις δυνατότητες να αποφέρουν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση αυτών των κοινωνικών ζητημάτων. Αυτά τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για κοινωνικά προγράμματα, και θα οδηγήσουν τις ε, κοινωνικές επιχειρήσεις να αποδείξουν το πόσο αποτελεσματικές είναι. Εσείς λοιπόν με ε, αυτή την υποστήριξή σας αυτής της πρωτοβουλίας μπορείτε να κάνετε μια πολύ μεγάλη διαφορά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην δεύτερη ομιλήτρια, τη Μίριαμ. Πριν um, Να κάνω σχόλια για τον κανονισμό. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το Ίδρυμα Schwab, που ήταν η πρώτη οργάνωση που υποστήριξε στην Ευρώπη τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Δημιουργήθηκε το 2000 από τον Κλάου Schwab, που δημιούργησε και το World Economic Forum και τη γυναίκα του, τη Hilde, εμείς πρέπει να πω ότι περνάμε από το μικροσκόπιο γύρω στις χίλιες κοινωνικές επιχειρήσεις και επιλέγουμε τελικά 25 με 30 ε, από τις επιχειρήσεις που παρουσιάζονται παγκοσμίων και σήμερα έχουμε 200 τέτοιους κοινωνικούς εταίρους δεν ε, παρέχουμε οικονομική υποστήριξη, αλλά διευκολύνουμε τις ε, διασυνδέσεις και τις επαφές με επενδυτές, με τις επιχειρήσεις, με το δημόσιο τομέα κτλ. Ε, και βεβαίως έχουμε πάντα εκ των υστέρων και το feedback όλων των επιχειρηματιών και αυτό είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε και ένα ε, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική καινοτομία, το πράγμα το οποίο είναι μέρος του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ και, της, ε, και των Συμβουλίων των σχετικών για θέματα που καλύπτουν τα περισσότερους τομείς που μας ενδιαφέρουν και πρέπει να πω ότι και ο κύριος Ντόναγιου ε, είναι μεταξύ αυτών των εμπειρογνωμόνων που είναι μέλος της τροπής αυτής. Αυτοί οι εμπειρογνώμονες με τη δουλειά τους και με βοήθησαν και με την δική μου εμπειρία τα τελευταία δέκα χρόνια να σας παρουσιάσω κάποια θέματα. Πρώτα απ' όλα, ποιος είναι ε, ο ορισμός αυτών των κοινωνικών επιχειρήσεων. Ένα θέμα θα αναφέρω. Τι κάνουν πρώτα απ' όλα οι, κοινωνικοί, οι επιχειρηματίες των κοινωνικών επιχειρήσεων. Πρώτα απ' όλα αφιερώνουν περίπου το 50% του χρόνου τους στο να μπορέσουν να αντλήσουν και να βρουν κεφάλαια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ευρεθούν τα χρήματα και επενδύσει που χρειάζονται. Ποια είναι, τι διαπιστώνουμε, ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο να βρουν επενδυτές που θέλουν να παρέχουν κεφάλαια ή δάνεια της τάξης των 200.000 έω 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός λοιπόν είναι ένας τομέα στον οποίο κάτι θα πρέπει να κάνουμε δεδομένου ότι θα πρέπει για να διευκολυθούν οι επενδύσεις στον τομέα αυτό να βρούμε και τα κατάλληλα κονδύλια και κεφάλαια από το δημόσιο τομέα. Υπάρχουν θέματα τα οποία κάλυψε ο συνάδελφος Ντόνεχιου και θα πρέπει να αναφέρω ότι πρώτα απ' όλα εκ μέρους των κοινωνικών επιχειρήσεων δεν υπάρχει εμπειρία στο να συλλέγουν ε, τα κονδύλια που χρειάζονται και ε, θα πρέπει επίσης να παρέχουν και τα κατάλληλα ε, κονδύλια ώστε να γίνεται η τεχνική βοήθεια και να μπορέσουν να βοηθήσουν μία επιχείρηση να σταθεί στα πόδια της από το πρώτο στάδιο. Επίσης θα πρέπει να βρούνε τους κατάλληλους μηχανισμούς ε, αναφοράς χωρίς να δημιουργήσουν υπερβολικό φόρτο με, στις, κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο θα πρέπει ως πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, ήδη έχουμε δει ε, τέτοιου είδους ε, στάντας, τέτοιου είδους ε, πρότυπα αναφοράς να δημιουργούνται στην αγορά και θα πρέπει στην ΕΣΜΑ να δούμε πώς, να δούμε πώς τα ταμεία αυτά θα αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα των προτύπων τα επόμενα χρόνια. Εάν υπάρχει μία βάση δεδομένων θα βοηθηθούν πάρα πολύ όλες οι επιχειρήσεις του τομέα πόσο σημαντικά είναι τα σήματα. Σε όποιον και αν μίλησα, λέγουν ότι θα χαιρετήσουν την ύπαρξη αυτού του ευρωπαϊκού σήματος. Τα χαρτοφυλάκια τους θα, τους επιτρέπουν, θα πρέπει να τους επιτρέπουν να κάνουν και επενδύσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι τα ποσοστά τα οποία θα πρέπει να επενδυθούν ώστε να θεωρηθεί ότι πρόκειται για επένδυση ε, με κοινωνικό αντίκτυπο. Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτά τα ποσοστά θα πρέπει να ανέβουν στο 80-90% ενώ θα πρέπει ο υπεύθυνο να διαθέτει και μια κάποια ρευστότητα. Αλλά περίπου το ποσοστό του 70% θεωρείται ένα καλό ποσοστό για να αρχίσει μια τέτοια επιχείρηση. Τελειώνοντα, θα ήθελα να πω ότι θα θέλαμε να υπάρχουν στην Ευρώπη δυνατότητες να μπορεί να κάνει την μέτρηση αυτών των ε, ε, ε, επενδύσεων, αν θέλετε, που έχουν μια κάποια κοινωνική αξία και σημασία. Πρώτα απ' όλα με την εισαγωγή φορολογικών κινήτρων, ώστε να μπορέσουν να ενθαρρυνθούν οι επενδυτές να επενδύσουν σε τέτοιου είδους κοινέ επιχειρήσεις και δεύτερον, να δοθούν ε, δυνατότητες να έχει κανείς μία μικρή απόδοση στο κεφάλαιο το οποίο επενδύεται και να υπάρχει και ε, σύμπραξη μεταξύ ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαν με τον τρόπο αυτό να δοθούν κίνητρα για να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις στον τομέα αυτό των κοινωνικών επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ που μας δώσετε την ευκαιρία να είμαστε και να σας εξηγήσουμε τις απόψεις μας. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι τώρα η διαδικασία θα είχε ως εξής. Στρέφομαι προς τα μέλη ή ε, μάλλον πρώτα θα απευθυνθώ στους κοιόδης γιατί έχουμε περιορισμούς χρόνου. Έτσι λοιπόν θα μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις και θα επανέλθουμε στους ομιλητές μας και τέλος τον εισηγητή. Μέλη, λοιπόν, αγαπητά μέλη, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις στους ομιλητές και μπορείτε να σχολιάσετε και το σχέδιο έκθεσης. Ε, ε, έρχομαι πρώτα στον Σαΐντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε δύο Σαΐντ λοιπόν εδώ πέρα όπως φαίνεται. Ε, μπερδεύτηκα κιόλας και με τον καφέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά και θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την εισηγήτρια και βεβαίως τους δύο εμπειρογνώμονες προσκεκλημένους μας. Θα ήθελα να πω το εξής. Έχω την εντύπωση ότι στα περισσότερα κράτη-μέλη αυτή η έννοια της κοινωνικής ε, οικονομίας είναι μια καινούρια έννοια και συνήθως αυτό είναι κάτι που το αναλαμβάνουν οι αρχές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Όμως, κάλλιστα μπορεί κανείς να δει και την παρουσία και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν συγκεκριμένες επενδύσεις ε, στην κοινωνική οικονομία από μέρους του ιδιωτικού τομέα και θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα ευρωπαϊκό σήμα στον τομέα αυτό. Ο ιδιωτικός τομέας σήμερα φαίνεται ότι επιθυμεί να αυξήσει τις κοινωνικά υπεύθυνες ε, επενδύσεις. Και θεωρώ ότι ένα ευρωπαϊκό σήμα καλύτερα θα μπορούσε να βοηθήσει όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις τους ή τις γνώσεις τους, υιοθετώντα και στηρίζοντας προγράμματα της κοινωνικής αυτής οικονομίας. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι χρειάζεται ένα καθεστώς ελαστικό, ευέλικτο, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών που θα ενδιαφερθούν ε, για αυτού του είδους τα προγράμματα. Υπάρχει εξάλλου και η περίπτωση κάποιων που θα επενδύσουν συλλογικά. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μήπως το ανώτατο όριο, μάλλον το κατώτατο όριο είναι πολύ υψηλό. Αυτή είναι μια ερώτηση που κάνω ε, και στους εισηγητές αλλά και στους εμπειρογνώμονες. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν ε, πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί ανάλογα με το κράτος μέλος, παραδείγματος χάρη, στο οποίο δίνεται ορισμός για το ποιος είναι ένας ε, κοινωνικός επενδυτής και τι ακριβώς είναι αυτά τα κοινωνικά προγράμματα θα εξαρτηθεί από το είδος, την κατηγορία του προγράμματος και ενδεχομένως θα υπάρχουν και κάποιες γκρίζες ζώνες μεταξύ της λεγόμενης πραγματικής οικονομίας και της κοινωνικής οικονομίας. Και αυτό θα ήθελα να μου απαντήσουν ε, οι εμπειρογνώμονες πώς το βλέπουν. Τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι πέρα από αυτό το διαβατήριο, αυτό το σήμα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι να επενδύσει κανείς ε, σε προγράμματα της κοινωνικής οικονομίας. Βεβαίως εδώ υπάρχει τελείως διαφορετική φορολογική πολιτική και διαφορετικοί κανόνες ε, για τη χρηματοδότηση. Μήπως θα μπορούσαμε εδώ να συντονίσουμε λίγο τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ όλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Εισηγήτρια για τις εισαγωγικές παρατηρήσεις σας. Ήθελα εγώ να κάνω την ίδια ερώτηση όσον αφορά τον ορισμό και όσον αφορά αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες ε, επαγγελματιών επενδυτών ή γενικών επενδυτών. Θα θέλαμε να μας αναλύσετε λίγο περισσότερο το 70% που αναφέρατε. Είναι ένα κατόφλιο ή πως θα έπρεπε να είναι περισσότερο ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Θα ήθελα να μου πείτε κάποια καλά παραδείγματα. Διάβασα μερικά από αυτά εδώ. Μπορώ να σας πω αφού ότι δεν πείθομαι και δεν με πείθει ούτε ο ορισμός. Μήπως θα μπορούσατε λοιπόν να μου δώσετε... Γιατί πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία εδώ πέρα. Εδώ πέρα και μετά χρειαζόμαστε επίσης και μια κοινωνική προστιθέμενη αξία. Εγώ δεν είμαι επαγγελματία. Είμαι ένας απλός επενδυτής. Ας πούμε. Και επενδύω σε πολλές τέτοιες ας πούμε κοινωνικές επιχειρήσεις ε, και ίσως δεν χρειάζομαι την απόδοση μόνο, χρειάζομαι κάτι παραπάνω, χρειάζομαι κάποια καλά παραδείγματα κάποια πιστικά παραδείγματα ώστε να είμαι βέβαιος ότι αυτοί οι οργανισμοί, αυτές οι εταιρείες παρέχουν αυτά που υπόσχονται. Και επίσης η τελευταία ερώτηση είναι θα μπορούσε να υπάρξει κατάχρηση σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις, αν το προσέξετε, κατάχρησης σε αυτές τις τράπεζες. Ευχαριστώ. Φίλιπ. Καταρχήν ε, είμαι ο Σβέν και θα σας απαντήσω γαλλικά για να με καταλάβει η Σοφή. Και εγώ θα ήθελα να κάνω κάποια θετικά σχόλια εξαιρετική εργασία. Πρόκειται για έναν τομέα πάρα πολύ σημαντικό, χρήσιμο, η κοινωνική οικονομία. Και είναι πολύ θετικό το ότι η Επιτροπή ενδιαφέρθηκε για το θέμα αυτό. Όσον αφορά την Επιτροπή της Σοφή, άρθρο 3. Η... χρησιμότητα να προσθεθούν εδώ κάποια άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Παραδείγματο χάρη να το θέμα του δανεισμού. Τροπολογία 32. Και αυτό συμβαδίζει με αυτά που είπε ο Σαΐντ. Δηλαδή το θέμα του μάρκετινγκ, των διαφόρων επενδυτικών ε, ταμείων, ιδιαίτερα των ατομικών επενδυτών. Και Βεβαίως οι διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή που θα πρέπει να συνοδεύουν αυτά τα μέτρα. Και ενώ υπάρχει αποταμίευση στην Ευρώπη, σκεφτείτε παραδείγματος χάρη την περίπτωση της κυβέρνησης του Βελγίου, μέσα σε μία εβδομάδα όταν ζητήθηκε η συνδρομή των, των Βέλγων πολιτών 5,6 δις, σχεδόν 6 δις μεταφέρθηκαν σε διάφορα προγράμματα. Και βεβαίως η απόδοση δεν είναι η μεγαλύτερη για τέτοιου είδους προγράμματα. Από την άλλη μεριά υπάρχει ε, σημαντικό απόθεμα στην αποταμίευση. Οι μικροεπενδυτές ενδεχομένως θα μπορούσαν να στραφούν προς τέτοιου είδους ε, προγράμματα. Τροπολογία 21. Εδώ συμφωνώ και εγώ ότι χρειάζονται κάποιοι δείκτες απόδοσης, οι οποίοι να είναι μετρήσιμοι. Άρθρο 3, κάπου θα πρέπει ίσως να πούμε πιο συγκεκριμένα τι είναι μια θετική κοινωνική, ένας θετικός κοινωνικός αντίκτυπος. Αν παραδείγματος χάρη θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας ένα ταμείο κοινωνικής, ε, κοινωνικών επενδύσεων που θα μπορούσε να βελτιώσει μια περιοχή η οποία έχει μολυνθεί, καταστραφεί από μια βιομηχανική δραστηριότητα. Και αυτό έχει ε, τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί στο κοινωνικό αντίκτυπο, το θετικό. Τροπολογία 33, ναι. Και εδώ μπορούμε να εν ενδυναμώσουμε τον ε, ρόλο της ΕΣΜΑ. Και Σοφή εδώ, ακούγοντας ε, τους δύο εμπειρογνώμονες, ε, θα συμφωνήσω μαζί τους και δεν έχω καμία συγκεκριμένη ερώτηση να κάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που διέκοψα πριν. Ε, πρέπει να σα εξηγήσουμε την λεπτή διαφορά μεταξύ Σαΐντ και Σάιντ. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον Νίκ και τη μου. Πολύ σημαντικό που ακούμε για τον αντίκτυπο μια τέτοια νομοθεσία. Ευχαριστούμε και την εισηγήτρια τη Σοφή επίση για αυτή τη συζήτηση. Πιστεύω ότι η ατμόσφαιρα αυτή τη συζήτηση είναι πολύ συνεργατική και είναι πολύ ενθαρρυντικό το να εργαζόμαστε σε ένα φάκελο με κοινού στόχους όλοι μαζί. Πραγματικά τίποτα δεν μας χωρίζει όσον αφορά τους στόχους που προσπαθούμε να επιτύχουμε στο πλαίσιο αυτού του φακέλου. Ε, δύο ερωτήσεις έχω να κάνω και δύο σχόλια. Από ό,τι κατάλαβα από τις συζητήσεις με την Κομισιόν γιατί θέλουν να περιοριστεί αυτό σε επαγγελματίες επενδυτές ώστε να οικοδομηθεί το σήμα και η φήμη είναι κρίμα που δεν μπορούμε να βρούμε ένα τρόπο. Θα ήθελα να μάθω πώς θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε και ιδιώτες επενδυτές ε, να γνωρίζουν τον κίνδυνο, να γνωρίζουν ότι, δεν, ότι αυτό στο οποίο επενδύουν είναι κοινωνική απόδοση και όχι οικονομική απαραίτητα, ώστε να επενδύσουν ε, με συνεργατικό τρόπο σε αυτά τα κοινωνικά συστήματα. Έχετε κάποια ιδέα γι' αυτό Δεύτερον, αναρωτιέμαι τι πιστεύετε όσον αφορά το κατόφλιο των 500 εκατομμυρίων και όσον αφορά το γεγονός ότι οι τιμές μπορεί να αυξομειώνονται καθημερινά, πώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό ρεαλιστικά. Κατά την άποψή σας υπάρχει λόγος να χάσουμε αυτό το σήμα και το τρίτο που θέλω να ρωτήσω, όσον αφορά τα ταμεία κοινωνική επιχειρηματικότητα, τι θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τη απέτηση ύπαρξη θεματοφύλακα, όπως την παρουσιάζει η συγγήτρια. Για εσά είναι μια θετική κίνηση, προσθέτει κάτι, έχει προσθέτω κόστο. εξαρτάται από κάποια πράγματα. Ήθελα να ακούσω τη δική σας απάντηση για το πόσο χρήσιμη είναι αυτή η απέτηση ύπαρξη θεματοφύλακα. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρος. Ο τελευταίος είναι ο Γιώργιον Κλούτερ. Υπάρχουν κάποια άλλα μέλη που θέλω να μιλήσω. Παρακαλώ να μου το αναφέρετε. Γιώργιον. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την έκθεση. Πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή βάση για την περαιτέρω συζήτηση. Θα ήθελα όμως να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συζήτηση, αυτή την ακρόαση για να ακουστούν κάποιες σημαντικές ε, ιδέες γύρω από τις οποίες θα πρέπει να σκεφτούμε, να συζητήσουμε, να επεξεργαστούμε και αυτό το κείμενο. Εργάζομαι εδώ και δεκαετίες ε, στον τομέα αυτό στη Γερμανία. Ξέρω πολύ καλά τον τομέα αυτό της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Και θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για έναν ε, τομέα, τουλάχιστον στη χώρα μου, ο οποίος ε, ουσιαστικά κατευθύνεται γύρω από τις ανάγκες ε, των ανθρώπων ε, και βεβαίως έχουμε μια σειρά συνοδευτικών μέτρων και πολιτικών όπως τη φορολογία που στρέφουν κάποιες επενδύσεις προς τον τομέα αυτό. Και αυτό βεβαίως στοχεύοντας κάποιες κατηγορίες, κάποιες κοινωνικές ομάδες. Θέλουμε κάθε φορά να κάνουμε μία ανάλυση του τι περιμένουν αυτές οι κοινωνικές ομάδες και αυτό βεβαίως σημαίνει κάθε φορά ότι ο τρόπος που λειτουργούν οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα πρέπει κάθε φορά να αλλάξει και πρέπει κάθε φορά να προσαρμοστούν στις ανάγκες. Και δεν ξέρουμε πάντα ποια είναι η κατεύθυνση. Υπάρχει πολλές φορές και μία συγκεκριμένη, αν θέλετε, απώλεια θα έλεγα. Εγώ έρχομαι στην Γερμανία από μία περιοχή η οποία είναι εξαιρετικά φτωχή. Χρειαζόμαστε λοιπόν να προσελκύσουμε χρήματα ιδιωτικούς, ε, αν θέλετε, πόρους σε μια περιοχή όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν υπάρχουν ε, άνθρωποι με δυνατότητες στην περιοχή αυτή. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε θέση να διαθέσουν επιπλέον πόρους. Και γι' αυτό και σας λέω ότι θα πρέπει να βρούμε αποτελεσματικά εργαλεία γιατί σε περιοχές όπως παραδείγματος χάνει το νότιο τμήμα της Γερμανίας όπου υπάρχουν ιδρύματα, υπάρχουν τρόποι χρηματοδότησης μέσω τέτοιων μορφών ε, κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το πρόβλημα είναι πολύ πιο ε, εύκολο να ξεπεραστεί, αλλά προβληματίζομαι για περιοχές όπως αυτήν από την οποία προέρχομαι. Εκεί είναι προβληματική η, αν θέλετε, προσέλκυση πόρων για τέτοιου είδους προγράμματα. Και δεν είναι εύκολο. Ε, γνωρίζω πολύ καλά ότι οι επενδυτές, αν θέλετε, έχουν πάρα πολλές επιλογές. Υπάρχει μεγάλος ενταγωνισμός όσον αφορά την ε, επενδυτική ικανότητα και ο ίδιος έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να στρέψω την προσοχή των επενδυτών παραδείγματο χάρη για τη δημιουργία κάποιων κέντρων για τους άνεργους είτε τη δημιουργία αν θέλετε πρωτοβουλειών για άτομα που ψάχνουν κάποιες δυνατότητες κατάρτισης. Δεν είναι τόσο ελκυστικά, αν θέλετε, τα προγράμματα αυτά για τους πιθανούς επενδυτές. Και εκεί είναι η δυσκολία. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Κανείς άλλος δεν έχει ζητήσει το λόγο. Προτείνω λοιπόν τώρα να επανέλθουμε στον Νίκ, τη Μυριάμ και μετά πάλι στη Σόφη. Έχουμε περίπου 15 λεπτά. Νίκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ να απαντήσω, να προσπαθήσω να απαντήσω μερικέ από αυτές τις ερωτήσει. Ε, μερικές από αυτές τι ακούσαμε πάνω από μία φορά. Η πρώτη ερώτηση είναι 100.000 υψηλότερο κατοφλό και αν χάνουμε κάτι. Κατά την άποψή μου, ναι. Υπάρχει βούληση σε κάθε επίπεδο και ακόμη σε μεγαλύτερο βαθμό ίσως από μικρούς επενδυτές. Το σκεπτικό είναι ότι ναι μεν υπάρχουν κίνδυνοι σε τέτοιου είδους επενδύσεις όπως σε κάθε επένδυση. Δεν πιστεύω ότι όταν μιλάμε για χρηματοδότηση δανειακή ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ε, ε, σε ε, επένδυση σε μια κοινωνική επιχείρηση από σε μια άλλη επιχείρηση. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι καλό θα ήταν να χαμηλώσουμε το όριο, το όριο εισόδου σε αυτά τα ταμεία. Όσον αφορά τον ορισμό, εδώ υπάρχει πρόβλημα σε ολόκληρο τον τομέα. Το κοινωνικό επιχειρηματικό κεφάλαιο το καθορίζουμε βάσει δύο χαρακτηριστικών. Το πρώτο είναι η κοινωνική αποστολή αυτή μπορεί να περιγραφεί από τον τρόπο των αποσχολούμενων ή την υπηρεσία που παρέχεται. Ωστόσο πρέπει να υπάρχει μια σαφώς καθορισμένη κοινωνική ε, αποστολή και να υπάρχει τα καταστατικά της επιχείρησης και δεύτερον τι κάνουν οι επιχειρήσεις με τα ε, κέρδη που αποκομίζουν και είναι σημαντικό να υπάρχει μια σαφής εικόνα είναι εύκολο σε ορισμένου οργανισμούς τύπου φιλανθρωπικούς οργανισμούς αλλά είναι πιο δύσκολο από όταν μιλάμε για κερδοφόρες επιχειρήσεις. Το πώς λοιπόν, ποια είναι η κοινωνική αποστολή, πώς ενσωματώνεται και τι γίνονται με τα κέρδη. Αυτά είναι τα ζητήματα. Αυτές είναι οι δύο κυριότερες ερωτήσεις στις οποίες ήθελα να απαντήσω. Κάποιος ανέφερε το ζήτημα της μάρκας, του σήματος, αν μπορεί να υπάρχει κατάχραση αυτού. Φυσικά, ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα, γι' αυτό απαιτείται σαφής έλεγχος και ορισμός του ποιο είναι επιλέξιμος και ποιε είναι οι επιλέξιμες επενδύσεις. Και χρειάζεται κάποια αριθμιστική παρακολούθηση όλων αυτών, επιτήρηση. Όλα αυτά καλύπτονται επίσης, ε, όπως αναφέρει και το έγγραφο, οι σαφείς ε, μετρήσεις ε, Όσον αφορά τα 500 εκατομμύρια ευρώ του κατοφλίου, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι απαραίτητο. Αυτό προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε είναι η κλίμακα στις κοινωνικές επιχειρήσεις ε, και στους οργανισμούς που τις διαχειρίζονται. Ευχαριστώ πολύ, Μίριαμ. Απλά ήθελα να προσθέσω σε όσα υπόθηκαν το όριο 100.000 για τους επενδυτές αυτό που είχαμε δει στον τομέα της μικροχρηματοδότησης που θεωρείται ότι βρίσκεται 10 χρόνια μπροστά στην περίπτωση των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι τα τελευταία χρόνια για παράδειγμα η Credit Suisse έχει ένα retail fund στο οποίο οι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν για μικροχρηματοδότηση Έχουμε την Κίβα που προέρχεται από τι ΗΠΑ η οποία παρέχει σε οποιονδήποτε μέσο διαδικτύου ένα πολύ απλό εργαλείο για την επένδυση έω και ενό ευρώ. Έχουμε λοιπόν ένα έτοιμο εργαλείο το οποίο μπορεί να μα δείξει το δρόμο για τον τομέα του retail fund. Θα έλεγα ότι τα μικρά ταμεία που υπάρχουν σήμερα στοχεύουν περίπου κουπόνια 100 ή παραπάνω, 100.000. Επειδή είναι αναποτελεσματικά τα υπόλοιπα. Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε σε χαμηλότερα tickets, ίσως και 50.000. Ακόμη και οι πλουσιότεροι του κόσμου θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο και που θα μπορούσαν να επενδύσουν ένα πολύ μικρό ποσοστό του χαρτοφυλακίου τους. 100.000 λοιπόν, αν είναι το 1% ε, των ρευστών που διαθέτει κάποιος, ε, ο ορισμός, ε, όπως είδαμε, ε, υπάρχει αυτή η γκρίζα ζώνη. Μπορεί να υπάρχει κινδύνος κατάχρησης διαφορετικών ερμηνεών αυτή τη στιγμή. Μαζί με τους δικούς μας κοινωνικούς επιχειρηματίες που γνωρίζουμε, προσπαθούμε να ορίσουμε το όριο μεταξύ κοινωνικής επιχείρησης και εμπορικής εταιρείας που μπορεί να είναι ε, υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Έχει σχέση με τις μορφές ιδιοκτησίας, με την κατανομή των κερδών, ίσως με τους υψηλότερους και τους χαμηλότερους μισθούς, τα ζητήματα διαφάνειας, διακυβέρνησης και έτσι βλέπουμε πολλές ε, επιπλέον πληροφορίες να προκύπτουν σε αυτό το πεδίο. Όσο αφορά την πιο γενική φιλοσοφική ερώτηση όσον αφορά τον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων, το πεδίο εφαρμογή των κοινωνικών επιχειρήσεων, και εγώ είμαι Γερμανίδα και γνωρίζω τη γερμανική συζήτηση που έχει γίνει για το Ευρω... γερμανικό κοινωνικό κράτο, οι κοινωνικοί επιχειρηματίε, όπω βλέπουμε, αποτελούν μια πολύτιμη προσθήκη στο υπάρχουσε δομέ κοινωνικού κράτου. Συνήθω έχουν πιο καινοτόμου και αποδοτικού μηχανισμού που συμπληρώνουν τι υπάρχουσε δομέ. Ο κοινωνικός επιχειρηματίας συνήθως προέρχεται από το υπάρχον περιβάλλον. Έτσι γνωρίζει ακριβώς τις ανάγκες των ανθρώπων, τις οποίες προσπαθεί να αντιμετωπίσει και συχνά ανακαλύπτουν αρκετά ικανούς μηχανισμούς για κάτι τέτοιο. Ε, ίσως είναι μεγάλη πρόκληση η έβρεση χρημάτων σε αυτούς τους τομείς. Ε, γι' αυτό βλέπουμε τέτοια ταμεία ξεκινούν σε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Μόναχο, η Γενέβη και η Ζηρίχη και όχι απαραίτητα ε, στην περιοχή ας πούμε του Ρουρ ε, αλλά θα αναζητήσουμε και ευκαιρίες στις ε, λιγότερο πλεονεκτούσες περιοχές. Πρέπει να δώσουμε περισσότερη τώρα έμφαση σε τοπικές επενδύσεις. Πολλά σε κοινωνικά ταμεία στη Γερμανία λένε ότι θέλουν να επενδύσουν μόνο σε γερμανόφωνες περιοχές διότι θέλουν να προσθέσουν αξία εκτός από χρήματα αυτό θεωρώ ότι δεν είναι μεγάλο πρόβλημα το να περιοριστούν αναγκαστικά σε απλά επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι βλέπουμε και έναν άλλο τύπο ταμείου που ξεκινάει να γίνεται βιομηχανία, όπου θα έχανε η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν περιόριζε τις ευκαιρίες επένδυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε τώρα ταμεία που βρίσκονται είτε στο Λουξεμβούργο είτε στην Ελβετία. Είναι ενδιαφέρουσε ιδέε όσον αφορά την οικοδόμηση μια μεγάλη βιομηχανία που θα είναι παγκόσμια. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Και η Σόφη έχει τώρα το λόγο. Σύντομα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ καταρχήν θεωρώ ότι η έκθεση αυτή εξελίσσεται σε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Η Επιτροπή πραγματικά έχει κάνει εξαιρετική εργασία και το κλίμα στο οποίο διεξάγεται αυτή η συζήτηση είναι σίγουρα αποτέλεσμα της εργασίας που έχει γίνει από την Επιτροπή. Ευχαριστώ τους σκιώδης ηγητές για την ανάλυση τους, τα σχόλιά τους. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Θα τις δούμε αργότερα. Όσον αφορά τώρα το να ανοίξει αυτό, αυτή η χρηματοδότηση και σε ιδιώτες, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιδέα. Την έχω σκεφτεί, πρέπει να την συζητήσουμε. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα, αν θέλετε, είναι κάτι καινούριο. Ίσως μπορεί να φανεί και επικίνδυνη η επένδυση. Και γι' αυτό και είχα σκεφτεί ότι ίσως προστατεύουμε τους ε, ε, επενδυτές ε, ιδιώτες, εάν για κάποια χρόνια δεν έχουν πρόσβαση καθότι είναι ίσως ακόμα λίγο επικίνδυνος ο τομέας. Αλλά βεβαίως μπορούμε να το συζητήσουμε. Τώρα για τις μεγάλες εταιρείες, το κατόφλι επίσης θα πρέπει να συζητηθεί. Θεωρώ ότι Καταρχήν έπρεπε να θέσουμε ένα όριο. Αλλά μπορούμε να επανεξετάσουμε και το αν μπορεί αυτή η επενδυτική δυνατότητα να ανοίξει και για τις μεγάλες εταιρείες αλλά και για τους ε, ιδιώτες. Κύριε Κλουτέ, είπατε ότι αυτό αφορά μόνο τις ε, επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, γιατί πρόκειται για έναν μοχλό Πρόκειται για επενδύσεις που μπορούν να οδηγήσουν, μπορεί να οδηγήσουν σε νέες θέσεις απασχόλησης. Γι' αυτό και είμαι υπέρ του να επωφεληθούν καταρχήν αυτές οι επενδύσεις, ε, να επωφεληθούν από αυτές τις επενδύσεις οι δικές μας επιχειρήσεις, τουλάχιστον καταρχήν. Ε, έχουμε ανάγκη να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτή ήταν η ιδέα μου καταρχήν. Και κάτι άλλο, αλλά υπάρχουν πολλές ε, ερωτήσεις, θα τις απαντήσω όλες. Το θέμα της προστασίας των επενδύσεων, διατηρώντας μια σχετική ελαστικότητα και βεβαίως έχοντας κάποιες εγγύσεις. Γι' αυτό και εγώ επέλεξα αυτή τη μέθοδο. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι ιδέες που ακούστηκαν. Ευχαριστώ άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία που πραγματικά μας συνοδεύει με πολύ ανοιχτό πνεύμα. Ευχαριστώ άλλη μια φορά όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση και βεβαίως ε, ιδιαίτερα ευχαριστώ τους ε, εμπειρογνώμονες. Thank ευχαριστώ. Θα ήθελα να περάσουμε αμέσως στο επόμενο θέμα, αλλά δεν μπορούμε να αρχίσουμε πριν από τις 4 και 4. Διότι ίσως κάποιοι σκιώδεις γιατί δεν είναι παρόντες. Για να δούμε. Η Ντανούτα Χούμπνερ δεν είναι εδώ, αλλά οι πρόεδροι των επιτροπών δεν μπορούν να απελευθερωθούν εύκολα. Θέλετε να αρχίσουμε μέσως, μπορούμε. Ας χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διαθέσή μας. Φιλίπ, σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Σάραν. Σας ευχαριστώ όλους τους Είμαι πρώτη φορά εισηγητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι εντυπωσιασμένο. Αλλά πάντα υπάρχει μια αρχή για όλα. Να είστε καλοί λοιπόν μαζί μου. Δεν πρόκειται βεβαίω για ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Αρχίζοντα, θα ήθελα να κάνω το... εξή Το 2008 είδα κάποια αποτελέσματα οι οποίες είχαν γίνει από κάποιες επιχειρήσεις επιχειρηματικού ε, κεφαλαίου και καινοτομίας από κάποιες επιχειρήσεις. Και είχα δει διάφορα στοιχεία τα πλαίσια του Green Tech. Και είχα δει ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης στον τομέα αυτό. Βεβαίως, η απάντηση στο πρόβλημα των αδυναμιών μας δεν είναι μόνο η ύπαρξη μιας ενός κανονισμού. Κυρίως είναι θέμα στάσεις των Ευρωπαίων που δεν είναι αρκετά τολμηροί, που δεν επιχειρούν, που δεν, και αν κάνουν λάθος ας ξαναρχίσουν. Μας λείπει αυτό το στοιχείο σε σχέση με τους Αμερικανούς στην Ευρώπη. Καλό είναι αυτό το κομμάτι της νομοθεσίας λοιπόν που εξετάζουμε, ώστε να μπορέσουν οι πάντες να είναι στην, ε, στην ίδια βάση. Καλό είναι αυτό και για τους ε, επενδυτές ε, στην Ευρώπη και κάποιοι μου είπαν μην πιστεύετε ότι θα έχετε επενδύσεις, μεγάλες επενδυτές σε όλη την Ευρώπη. Εδώ έχουμε να κάνουμε κυρίως με τέτοιους επιχειρήσεις τις οποίες επενδύουν μικροί ε, επιχειρηματίες. Όπως και η Σοφή, έκανα και εγώ κάποιες ε, αλλαγές και μπορούμε να συζητήσουμε κάποια θέματα. Εγώ λέγω κάποια πράγματα όσον αφορά τον ορισμό που των ε, εταιριών επιχειρηματικού κεφαλαίου, όσον αφορά την έδρα τους. Επίσης αυτό το οποίο λέγεται στο κείμενο είναι ότι δεν θέλουμε να ληφθούν υπόψη ε, τα επιχειρηματικά κεφάλαια τα οποία δραστηριοποιούνται σε φορολογικούς ε, παραδείσους. Αυτούς δεν θα πρέπει να δοθεί το περίφημο σήμα. Επίσης αυτό το οποίο θα ήθελα είναι να μπορούν ε, να γίνονται επενδύσεις από μια τέτοιου είδους εταιρεία σε μία άλλη και θα πρέπει επίσης ε, να δούμε πόσο λαμβάνουν υπόψη οι επιχειρηματίες τέτοιου επιχειρήσεων τους ε, ε, εργαζομένους τους για να τους προστατεύσουμε βάσει του κοινοτικού δικαίου. Τώρα, σαν αφορά την δαφάνεια που θα πρέπει να ισχύει από τέτοιου είδους εταιρείες, επίσης αναφέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, η βασική πρόταση της Επιτροπής πρέπει να πω ότι δεν ήταν πάρα πολύ πολύπλοκη άμα νομοθετικής ε, πλευράς και εν περιπτώσει πρόκειται για την πρώτη εξέταση τώρα του θέματος αυτούς. Τώρα, θα δείτε από τον αριθμό των ατόμων, από το, τα άτομα που χειρίζονται μάλλον αυτό το φάκελο, ότι πρόκειται για ένα βελγικό φάκελο. Μας αφορά εμάς το Βέλγιο, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε ανοιχτοί όμως ξέρετε στο Βέλγιο και δεχόμαστε παρατηρήσεις και υποδείξεις από τον οποιοδήποτε. Ακόμη και η Σουηδή, η Γερμανία, οποιοδήποτε άλλο θέλει να κάνει παρατηρήσει είναι καλοδεχούμενος. Ευχαριστούμε. Αν έχουμε και από τους συναδέλφους του Ηνωμένου Βασιλείου κάποιες ε, ή ε, από από το Ηνωμένο Βασίλειο κάποιες υποδείξεις και παρατηρήσεις και αυτές καλόδεχτες είναι γιατί εσείς έχετε μία διαφορετική νομοτροπία και δεν θα πρέπει ότι προέρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία να το αγνοούμε. Και εσείς ισότιμοι εμά είστε. Κάντε μας, κάντε τι προτάσεις. Για πρώτη φορά όμω θα πρέπει να πω ότι Νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ Πρασίνων και ε, Βρετανών, αν θέλετε. Και θα δούμε που θα καταλήξει. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε έτσι που συμφωνείτε. Δίνουμε το λόγο τώρα σε δύο μιλητές ε, για το θέμα αυτό. Έχουμε τον Τζος Πίτερς managing partner της Capricorn Venture Partners και με την ε, καθηγήτρια Sophie Menegard της GIMV Private Equity είναι πρόεδρος έχετε ε, τα βιογραφικά τους ε, αν δεν έχετε αντίρρηση Μπορείτε να μιλήσετε με αυτή τη σειρά. Τζο, λοιπόν, πρώτο. Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις απόψει μου και να απαντήσω σε οποιασδήποτε απορίες μπορείτε να έχετε για το κατά πόσα η πρόταση για τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου της Κομισιόν είναι επαρκής για να κινητοποιήσει τη βιομηχανία επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ευρώπη και να προέχει πρόσβαση σε equity finance και πώς θα μπορούσε το προτινόμενο καθεστώς να υλοποιηθεί πρακτικά. Θα βασίσω τα σύντομα σχόλια μου στην εμπειρία μου που είναι εδώ και πάνω από 26 χρόνια. Ε, υπήρξα πρόεδρος το 89-90 της Joint Venture Capital Association και ενεπλάκην στη δημιουργία της ISTAC ε, χρηματιστηρίου για τις ε, υποανάπτυξη εταιρείε στην Ευρώπη. Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια βρισκόμαστε στη Capricorn Virtue Partners εδώ στη Λουβένη του Βελγίου. Έχουμε ε, καταφέρει να βρούμε 150, πάνω από 150.000 ευρώ για επενδύσεις σε ε, επιχειρήσεις καθαρών τεχνολογιών και ε, τεχνολογικών υγείας στη Φιλανδία, στο Λουξεμβούργο, Έχουμε επενδύσει το μισό από αυτόν το ποσά σε 18 ευρωπαϊκές ΜΜΕ και σε 9 ευρωπαϊκές χώρες. μετά από τη συμπερίληψη των κεφαλών επιχειρηματικού κινδύνου στην οδηγία FIMD πραγματικά Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε την ανάγκη για ένα συγκεκριμένο καθεστώ για τα επιχειρηματικά κεφάλαια, πιο ευθυγραμμισμένο με το μέγεθο των ταμείων ε, επιχειρηματικών κεφαλαίων και με την έλλειψη συστημικών κινδύνων ε, με την οικονομική του σπουδαιότητα για τη χρηματοδότηση της καινοτόμου ανάπτυξης και των σχετικών ΜΜΕ και το ρόλο τους ε, για τη δημιουργία αποτελεσμάτων όπως δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη, σημαντικών επενδύσεων στην Ευρώπη, στην έρευνα και την ανάπτυξη. Είναι πως οποιαδήποτε πρωτοβουλία που μπορεί να, να οδηγήσει σε περισσότερη διάθεση επιχειρηματικού κεφαλαίου θα πρέπει να υποστηριχθεί. Ωστόσο πιστεύω ότι η βιομηχανία ευρωπαϊκών επιχειρηματικών κεφαλαίων έχει να αντιμετωπίσει σήμερα προκλήσεις που δεν φαίνεται να μπορούν να επιληθούν με ένα νέο ρυθμιστικό καθεστώς. Σήμερα ζούμε μία υπαρξιακή κρίση στη βιομηχανία μας. Τα τελευταία μεγέθη που δημοσιεύτηκαν την τελευταία εβδομάδα ε, από την ΕΦΚΑ στη Γενέβη δείχνουν ότι το 2011 ε, το συνολικό ποσό για επιχειρηματικό κεφαλαίων στην Ευρώπη που βρέθηκε ήταν 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήταν το 2 τρίτα του ποσού σε σχέση με το 89-90 όταν εγώ ήμουν πρόεδρος της ΕΦΚΑ ήταν μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό στι Ηνωμένε Πολιτείε. Πριν από μερικά χρόνια, ένα φοιτητή του MIT ε, συμπέρανε ότι η Ευρώπη δεν προσφέρει αρκετά χρήματα στι νοσίστατε επιχειρήσει του, οι οποίε, ωστόσο είναι κρίσιμε για τη μελλοντική ανάπτυξη και ευημερία και οι οποίες πρέπει να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιες αγοράς ε, με, παρκο... με ανεπαρκείς πόρους. Οι πρόσφατες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη, όπως το Φερεγγιώτα 2 και το Βασιλεία 3, έκαναν επενδύσεις ε, από αντίστοιχα ασφαλιστικές εταιρείες απαγορευτικά ακριβές σε σχέση με τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Για παράδειγμα, μια επένδυση σε ένα ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων που θα επενδύσει σε 10 ή 20 υποκειμενές εταιρείε ε, για, μια, για μια τέτοια επένδυση μια ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να θέσει στην άκρη το 50% του κεφαλαίου της ως ιδία κεφαλαία. Για επένδυση σε κρατικά ομόλογα η απέτηση κεφαλαίου είναι μηδενική η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών προβλέπει ότι οι κανόνες του Ισφαιρεγγιώτας 2 θα μεταβιβάσουν τις επενδύσεις από εταιρείε και μακροπρόθεσμα κεφαλαιακά έργα σε προϊόντα σταθερών εσόδων όπως τα ομόλογα. Έτσι λοιπόν οι συστημικοί ε, κίνδυνοι θα αυξηθούν αντί να μειωθούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος οι ίδιες κεφαλαίκες απαιτήσει του Ισφαιρεγγιώτας 2 να εφαρμοστούν σε του ταμεία ε, όσον αφορά την οδηγία EORP. Όταν θα υλοποιηθεί θα έχει ως αποτέλεσμα μια άλλη κατηγορία επενδυτών οι οποίοι λόγω των ρυθμίσεων θα αποφεύγουν να επενδύουν σε ταμεία ε, επιχειρηματικών κεφαλαίων. Συμπέρανω λοιπόν ότι η πρόταση της Κομισιόν για τη ρύθμιση των EVCF είναι ενδιαφέρουσα αλλά είναι απίθανο να είναι επαρκής ε, για να δώσει επαρκή όθηση στη βιομηχανία ευρωπαϊκών επιχειρηματικών κεφαλαίων. Πολλές ε, πρόσφατα ε, πολύ πρόσφατα υιοθετηθέντες κανονισμοί και επηρεάζουν αρνητικά τη βιομηχανία μας και θα πρέπει να δώσετε προσοχή εάν θέλετε να επιτύχετε το στόχο σα για την ενίσχυση τη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση στην Ευρώπη. Όσον αφορά το κατά πόσο ο προτινόμενο κανονισμό είναι κατάλληλο, δεν θα κάνω οποιαδήποτε κρίση πριν από τη λεπτομερή υλοποίηση αυτού του καθεστώτας. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε το φόρτο για το καθεστώς αυτό των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών κεφαλαίων όσο το δυνατόν πιο ελαφρύ. Κατά την απόψή μου πρέπει να επιτύχουμε μια σωστή ισορροπία σε θέματα πεδίου εφαρμογή και φόρτου όσον αφορά το καθεστώ για τα ευρωπαϊκά επιχειρηματικά κεφάλαια. Εάν το πεδίο εφαρμογή είναι υπερβολικό στενό, κανεί δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει το διαβατήριο. Ο στόχο διευκόλυνση ε, τη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα εκπληρωθεί. Εάν ο Φόρτο είναι υπερβολικά υψηλό ε, για του αντίστοιχου μάνατζερ δεν θα υπάρχει κανένα πλέον έκτημα για τη χρήση του σήματος αυτού του καθεστώτος. Οι επιπτώσεις στο Φερεγγιώτα 2, της Βασιλείας 3, υπό το νέο καθεστώς ε, δεν θα βρίσκονται καθόλου εύκολα χρήματα για τέτοια επιχειρηματικά κεφάλαια. Ευχαριστώ πολύ και είμαι διαθέσιμος να απαντήσω τι ερωτήσει σα. Ευχαριστώ πολύ αρκετά μέλη αυτή τη επιτροπή. Ε, Θέλω να κάνω ερωτήσεις σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το equity. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε για τη φερεγγιότητα. Περνάμε τώρα στη Σόφη. Good uh, Χαίρετε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε να σας μιλήσω για την πρόταση αυτής της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τις αρχικές παρατηρήσεις που έγιναν ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα στην Ευρώπη να υποστηρίξουμε πλήρως τις καινοτόμες ΜΜΕ. Πρέπει να σας πω ότι εγώ έκανα την παρέμβασή μου, τον προετοίμασα πριν να δω Ποιε είναι οι τροπολογίε που έχουν κατατεθεί. τι είδα Και κάποιοι από τους φόβους που εκφράζω εδώ πέρα ε, δεν ισχύουν πλέον. Έχουν απαντηθεί κάποια ερωτήματα, γι' αυτό δεν θα τα επαναλαμβάνω. Τώρα, εάν η πρόταση αυτή θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις αυτές επιχειρηματικού κεφαλαίου, συμφωνώ και εγώ με τον Ζώσο ότι υπάρχουν πιο αρνητικά παρά θετικά σημεία τα οποία απορρέουν από αυτή την πρόταση. Αλλά είναι καλή ιδέα να έχουμε ένα καλό σήμα στις αγορές με, για αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν θα κάνει κακό. Εάν όντως εφαρμοστεί σωστά η οδηγία και δεν δημιουργήσει μεγάλο άχθος για αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει τέτοιου είδους επιχειρηματικού κεφαλαίου εταιρείε γίνει το χειροκροτούμε. Ό,τι δημιουργεί πρόβλημα να το, να το αποφύγουμε. Τέτοιου είδους εταιρείε πρέπει να πω ότι είναι πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες στη ΣΥΠΑ, άρα οι φιλοδοξίες τους, αν θέλετε, είναι περιορισμένες εμβέλεια σε σχέση με τον υπολείπων. Αν θα λυθούν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα αυτό, όχι. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η χρηματοδότηση αυτών των εταιριών επιχειρηματικού κεφαλαίου αφορά μόνο ένα πολύ μικρό μέρος εταιριών. Ακόμη και για τις καινοτόμες εταιρείες όταν μιλάμε ή για αυτές οι οποίες είναι αναπτυξιακές. Αυτή λοιπόν το μικρό ποσοστό εταιριών στις, ε, ακόμη και στη ΣΥΠΑ που μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια είναι πάρα πολύ μικρές. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αν λυθεί αυτό το πρόβλημα θα λυθούν όλα τα προβλήματα και φερεγγυότητας που έχουν αυτές οι περισκευστότητες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που βοηθάνε, αυτοί οι άγγελοι των επιχειρήσεων που λέγονται, οι οποίοι βοηθούν πολύ περισσότερο ε, από ότι άλλου είδους προτάσεις, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης. Για να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε τέτοιου είδου επιχειρήσει, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μια πολύ καλή και ομαλή βετάβαση από ένα είδο επιχειρήσεω σε άλλο, ξέροντα ότι οι διάφορε εταιρείε, ανάλογα με τον τύπο του, χρειάζονται και διαφορετικέ επενδύσει, διαφορετικού τύπου επενδύσει. Αν τώρα λοιπόν εστιαστούμε μόνο σε εταιρείε επιχειρηματικού κεφαλαίου, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Και υποστηρίζω και αυτά που είπε και ο Ζωάς, ότι όντω υπάρχουν και άλλα θέματα στην Ευρώπη τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε διότι μπορούν να θέσουν εν κινδύνο τέτοιου είδου εταιρείε. Πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το καθεστώς στην πράξη, φαίνεται ότι το πρωταρχικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το εξής. Εάν δεν γίνει σωστή εφαρμογή των κανόνων, δεν θα υποβάλουν ε, ε, η αίτηση για να αποκτήσουν αυτό το σήμα πάρα πολλές εταιρείες, αλλά θα είναι κενό περιεχομένου ότι γίνει. Και θα πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα τι είδους ε, κεφάλαια τέτοιου είδους αν θέλετε μπορούν να είναι επιλέξιμα βάσει ποιων κανόνων. Δεύτερον, πώς θα πρέπει όταν ε, αποκτήσει κάποιος αυτό το διαβατήριο να συμπεριφερθεί και να ανταποκριθεί στον διοικητικό φόρτο. Επίσης, θα πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει επένδυση που πληρεί τις προϋποθέσεις. Στις τροπολογίες διάβασα ότι οι επενδύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να περιορίζονται σε επιχειρήσεις που ε, υπάρχουν εδώ και μία πενταετία μόνο, μου φαίνεται τρομερό αυτό. Δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί έχετε αυτό το κατόφλι της πενταετίας. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες αναπτύσσονται πλήρως και δραστηριοποιούνται πλήρως μετά μία πενταετία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν ε, πάρα πολύ αρμονικά. Δεύτερον, γιατί όταν μιλούμε για επενδύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, μιλούμε μόνο για το ίδιο κεφάλαιο, για αυτές τις ε, επιχειρήσεις. Πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλοί ε, είναι οι επιχειρηματίες που επενδύουν τα κεφάλαιά τους με τρόπο ειδικό ανάλογα με την φορολογική νομοθεσία και αν φύγει αυτή η έννοια του subordinated debt, νομίζω ότι δεν θα δώσουμε καμία ευκαιρία σε αυτές τις εταιρείες να αναπτυχθούν. Επίσης, νομίζω ότι εδώ αναφέρεται ότι οι επενδύσει που πληρούν τις προϋποθέσεις περιορίζονται μόνο σε μέσα τα οποία εκδίδουν οι εταιρείε χαρτοφυλακίου. Ίσως θα μπορούσαμε εδώ να σκεφτούμε την δυνατότητα ε, τα κεφάλαια της εταιρεία αυτού του τύπου επιχειρηματικού κεφαλαίου να τα αναλάβει κάποιος τη στιγμή που αρχίζει σιγά σιγά να, να αποχωρεί ο επιχειρηματίας άγγελος όπως λέγεται. Και τέλος, ποιοι είναι επίσης αυτοί οι επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις. Μου φαίνεται ότι και πάλι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι περιοριστικό και εδώ προβλέπεται ένα, ε, κατά το τόριο ένα όριο 100.000 ευρώ που νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Αν δει κανεί τι προτείνεται στις τροπολογίες όσον αφορά το άγχος, κυρίως όταν γίνεται λόγος για τους ε, επιχειρηματίες ε, ε, όλοι αυτοί οι ορισμοί που συμπεριλαμβάνονται εδώ είναι κάτι το οποίο είναι περιοριστικό και θα αποκλείσει πολλούς και γιατί εδώ γίνεται λόγος για πράσινες παιδίες και τροπολογίες. Νομίζω ότι είναι άσχετο αυτό. Επίσης θέλω να πω ότι οι εταιρείε επιχειρηματικού και φαλαίου εάν εστιαστούν μόνο σε πράσινες επενδύσεις και πάλι θα αποτελέσουν κάτι το πολύ περιοριστικό. Αυτά είχα να πω. Φιλίπ, θέλεις να πάρεις το λόγο. Ναι, ακούγοντας αυτά που είπατε, δηλαδή ότι αυτή η πρόταση είναι σχετικά καλή, αλλά ότι υπάρχουν άλλα νομοθετικά κείμενα, τα οποία ε, περιέχουν δυσκολίες. Ε, είναι λίγο αργά όμως, γιατί ψηφίζουμε αύριο. Το θέμα έχει προχωρήσει. Αν έχετε πολύ συγκεκριμένα σχόλια για κάποια τμήματα αυτών των νομοθετικών κειμένων που σας δημιουργούν πρόβλημα, θα ήθελα να το ακούσω. Just, Θέλετε να απαντήσετε τώρα. Αλλιώ έχουμε και τον ε, εισηγητή, τον Ότμαρ, ο οποίος ήρθε. Δεν ξέρω αν ε, θεωρείτε ότι αυτή η αρνητική κριτική είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Το θέμα του Solvency 2, το οποίο βεβαίως αναφέρεται στην έκθεσή σας. Πολύ σύντομα, Τζος. Όσον αφορά τις ανησυχίες από τη μεριά του επιχειρηματικού κεφαλαίου. Θα ήθελα να πω ότι βεβαίως και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά όταν κάποιος κάνει μια άμεση επένδυση σε μια ασφαλιστική, παραδείγματος χάρη, και σε μια συγκεκριμένη εταιρεία η οποία δεν είναι συγμένη, Υπάρχουν ε, τρόποι κατανομής αυτών των κεφαλαίων, παραδείγματος χάρη αν τα κατανείμετε σε 20 διαφορετικές εταιρείες, φυσικά και ο κίνδυνος ε, μοιράζεται αντίστοιχα. Και οι ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιαίτερα αυτές που ασφαλίζουν ε, τέτοιου είδους κινδύνους, έχουν μεγάλη, αν θέλετε, ανησυχία όσον αφορά την ασφάλιση τέτοιων ε, επενδύσεων και γι' αυτό και όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται και στη Βασιλεία 3 αλλά και στο Solvency 2 που αναφέρεται ιδιαίτερα στις ασφαλιστικές εταιρείες και αν κοιτάξετε τα στατιστικά στοιχεία τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη θα δείτε ότι οι τράπεζε είναι αυτέ, ο τραπεζικό τομέα, είναι αυτό που έχει συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην χρηματοδότηση των ε, κεφαλαίων τέτοιου είδου για τις ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις. Και όλα αυτά, αν τυχόν ε, εφαρμοστεί και τεθεί σε ισχύ ακριβώς το Solvency 2, θα είναι πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα για τέτοιου είδους επενδύσεις, για επενδύσεις σε τέτοιου είδους εταιρείε. Όπως ξέρετε, όταν αναφερόμαστε στα συνταξιοδοτικά ταμεία, στα ασφαλιστικά ταμεία, πρόκειται για πάρα πολύ μακροχρόνιες απαιτήσει. Και η ολοκλήρωση, παραδείγματος χάρη αυτών των επενδύσεων, η οποία είναι μια επένδυση πολλών ετών και η οποία σε αυτές τις περιπτώσεις ανταποκρίνεται και με τις διάφορες υποχρεώσεις των συνταξιοδοτικών αυτών ταμείων, των ασφαλιστικών αυτών ταμείων. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη υποχρέωση που έχουν αναλάβει τα ταμεία έναντι των δικαιούχων, των συνταξιούχων. Όλα αυτά επιβαρύνουν, αν θέλετε, τις ε, επενδύσεις σε αυτό το τομέα στην Ευρώπη και αυτό είναι και αν θέλετε, μία από τις τρεις βασικές ανησυχίες μας. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε που το κόμμα αυτό που μια ανεξάρτητη πηγή. Δεν ούτε ήθελε τώρα τον λόγο. Uh, thank you uh, very much. Ευχαριστώ πολύ, Σαρών. Είμαι σκιώδη συγγήτρια του ΕΛΚ, κοιτώντα τώρα τον κατάλογο των σκιωδών εισηγητών και των συναδέλφων σήμερα. Ζητώ συγγνώμη που δεν είμαι Βελγίδα. Αν θέλετε όμως να μου δώσετε την υπηκότητα, είναι ευπρόσδεκτη. Για να μιλήσω τώρα, για να σοβαρευτούμε λίγο, συμφωνώ με όσους λένε ότι αυτός ο κανονισμός είναι σημαντικός. Αποτελεί ένα βήμα μπροστά προς ε, έναν σοφά μια σοφά αγορά στην Ευρώπη. Η πρόκληση είναι να δούμε κατά πόσο αυτός ο κανονισμός συμβάλλει πραγματικά στην πιο σημαντική πρόκληση της Ευρώπης σήμερα την ανάπτυξη, τη δημιουργία ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν δεν αφορά μόνο να φροντίσουμε ο κανονισμός να μην βλάψει τη βιομηχανία, αλλά να τονώσει και την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Αυτή, αυτό είναι το καθήκον μας γενικά. Θα έλεγα ότι ο κανονισμός είναι ικανοποιητικός, αλλά φυσικά προκύπτουν ερωτήσεις για όλους μας βάσει των που, πληροφοριών που έχουμε λάβει. Ήθελα λοιπόν να αναφέρω μία ή δύο ερωτήσεις προς τους ε, ομιλητές μας για να μας διαφωτίσουν. Ένα από τα ζητήματα σχετίζεται με το γεγονός νομίζω το άρθρο 3D της πρότασης αναφέρει ότι δεν πρέπει να αναφέρονται qualified portfolios. Η ερώτηση μου είναι υπάρχει λόγος ε, οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε αυτές τις αγορές ανάπτυξη να μην περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κανονισμό. Η δεύτερη μου αμφιβολία αφορά αυτό που αναφέρθηκε ήδη αυτή την επένδυση των 100.000 χρειάζεται να είναι τόσο υψηλό αυτό το ποσό για να προσελκύσει μόνο επαγγελματίες επενδυτές. Μήπως κάποιο χαμηλότερο όριο 50.000, μήπως αυτό θα παρήχε παρόλα αυτά επαρχή διασφάλιση ότι θα υπάρχουν επαγγελματίες επενδυτές αλλά ταυτόχρονα δεν θα μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό των επενδυτών που θα ήθελαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη στην Ευρώπη. δεύτερη ερώτηση σχετίζεται με αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ ε, για τη σήμα. Θεωρείται ότι υπάρχει επαρκής αιτιολογία ε, για να υπάρχουν επιχειρηματικά κεφάλαια με πάνω από 500 εκατομμύρια. Μετά προς τον Φίλιπ Λαμπέρτς ε, επειδή συμμερίζομαι ορισμένες από τις τροπολογίες σας, ε, ειδικότερα όταν μιλάτε για την ανάγκη ε, σας υποστηρίζω, αλλά έχω δύο αμφιβολίες όμως εδώ. Η τροπολογία 13, όπου προτείνεται να περιοριζόμαστε σε εταιρείε νεότερες των 5 ετών. Όλοι γνωρίζουμε ωστόσο κάποια επιχείρηση που δεν είναι νεοσύστατη αλλά έχει ίδιες ανάγκες ανάπτυξης βάσει επενδύσεων που απαιτούν επιχειρηματικά κεφάλαια. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να εφαρμόσουμε και αυτή τη λύση και μετά το θέμα του θεματοφύλακα. Από όσο καταλαβαίνω στις χρηματαγορές και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το ζήτημα των θεματοφυλάκων. Εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία στα οποία θα επενδύουν τα ταμεία αυτά δεν είναι εισηγμένα. Τι ρολό θα παίζει λοιπόν ο θεματοφύλακας ενώ σαφέστατα θα αποτελούσε φόρτο. Θεωρώ ότι θα έπρεπε κάποιο να μας εξηγήσει πόσο μεγάλο θα είναι αυτό ο φόρτος. Και εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο έχω κάποια αμφιβολία όσον αφορά τις τροπολογίες. Ευχαριστώ Σάρων, ευχαριστώ. Ο Σάιν τώρα. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω τον κύριο Λάμπερ για την εξαιρετική του συνεργασία και την προσέγγιση του. Ευχαριστώ επίση και του δύο μιλητέ για την πολύ ενδιαφέρουσα και ανοιχτή συνομιλία και το διάλογο. Συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας πρέπει να βρούμε τρόπους τόνωσης των επενδύσεων σε καινοτόμες εταιρείε. Η πρόταση αυτή είναι καλή. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτό αρκεί, κατά πόσο μπορούμε να το βελτιώσουμε και ποια είναι η σχέση με άλλες νομοθεσίες και ποιες είναι οι συνέπειες άλλων νομοθεσιών που εμπλέκονται σε αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να πούμε κάτι γι' αυτό στην έκθεση. Υπάρχουν νομοθετικές πτυχές και προσεγγίσεις που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε. Θα σκεφτούμε το CRD4 για παράδειγμα και κάποιες άλλες νομοθετικές πράξεις. Επίση, υπάρχει και πια σύνδεση με πράγματα για τα οποία δεν έχουμε ακόμη μιλήσει. Σκεφτούμε το Horizon 2020, για παράδειγμα. Αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της παρούσας επιτροπής βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι η πρόταση της Κομισιόν θα μπορούσε να εστιαστεί στη περίοδο 2014-2020 όπου πολλά δισεκατομμύρια ευρώ μπορεί να διατεθούν ε, για τόνωση των επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε εδώ μια σύνδεση, έναν συσχετισμό. Αυτό το θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των χρημάτων των επενδυτών, που επενδύουν οι επενδυτές σε τέτοιου έργα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει μια καλή συσχέτιση μεταξύ της διαφάνειας και των θεμητού ανταγωνισμού, αλλά δεν θα πρέπει να τρομάξουμε και τους πιθανούς επενδυτές. Πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε μια ισορροπία. Επίσης υπάρχει το ζήτημα του ενιαίου θεματοφύλακα, το οποίο πρέπει να έχουμε στο νου μας. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια ισορροπία και θα ήθελα να μου πούν οι ομιλητέ τι πιστεύουν για αυτό το ζήτημα. Δεν πρέπει να, η προσέγγιση μας δεν πρέπει να είναι υπερβολικά περιοριστική. Περιορίζοντας το όλο αυτό σε εταιρείε ε, ηλικία έως 5 ετών. Δεν είμαι βέβαιος γιατί γίνεται αυτό. Φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιος λόγος. Επίσης το σχόλιο που ακούσαμε ε, σε σχέση με τους business angels ήταν πολύ ενδιαφέρον και τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει αν λέμε ότι τα ταμεία μπορούν να επενδύουν μόνο σε νέες ε, μετοχές. Αυτό θα δυσχαίραινε το έργο των business angels. Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω την εισηγήτρια. Αυτό αυτή η συζήτηση για τα, τα κλειστού και ανοιχτού τύπου τα open-ended και closed-ended. Δεν έχω καταλήξει κάποιο συμπέρασμα, αλλά από ό,τι κατάλαβα το closed-end fund, το ταμείο κλειστού τύπου, έχει κάποιο όριο και εισαγαγεί κάποιο είδου προθεσμία. Παρότι σε ορισμένε περιπτώσει ε, επενδύει κανείς σε μια εταιρεία και αυτή αρχίζει να αναπτύσσεται κατά την ορίμανση του Ταμείου. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερο κεφάλαιο κατά την περίοδο ανάπτυξή τη για να περάσει το επόμενο επίπεδο. Εάν το Ταμείο λοιπόν σταματήσει τη δραστηριότητά του εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, μπορεί η κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. σω χρειαζόμαστε λοιπόν μεγαλύτερη ευελιξία σε αυτό το θέμα χωρίς να περάσουμε φυσικά σε ένα εντελώς ανοιχτού τύπου ταμείο, θα πρέπει να υπάρχει κάποια μέση λύση. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω αφορά τη σχέση με τα δημοσία ευρωπαϊκά ταμεία. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο που σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να δώσουμε κάποια όθηση σε αυτό το διαβατήριο και να αρχίσουν τα πράγματα να κινούνται, ίσως θα έπρεπε να πούμε ότι όσον αφορά αυτά τα επίσημα ταμεία στα οποία συμμετέχει η Ευρώπη, Αυτά επίσης θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαβατήριο. Αυτό θα μπορούσε να προσελκύσει, να ελκύσει και τα υπόλοιπα ταμεία να πράξουν το ίδιο. Και έτσι οι άνθρωποι μπορεί να αρχίσουν να τα χρησιμοποιούν τώρα. Όσον αφορά το κατόφυλλο των 100.000 ευρώ, αυτό ίσως είναι λιγότερο σημαντικό από ότι για τα κοινωνικά ταμεία, ωστόσο θεωρώ ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε μια σωστή ισορροπία μεταξύ ε, της πλήρους απελευθέρωσης αυτού και από την άλλη της προστασίας των ιδιωτών επενδυτών. Θα έπρεπε επίσης να εξετάσουμε τα feeder funds, ε, τα οποία είναι ταμεία που συγκεντρώνουν χρήματα ε, για μικρούς επενδυτές. Φεντέρ, τα θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο του να ανοίξουμε αυτά τα ταμεία σε, μεγαλύτερη, σε ευρύτερη ομάδα στόχο με σωστές διασφαλίσεις και πρότυπα. Θα ολοκληρώνω εδώ. Φίλιπ, παρακαλώ. from this Belgium, uh, uh, a big thank you to, the rapporteur for the... Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα σχόλια. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τους δύο προσκεκλημένους μας και αυτά που ακούσαμε σαφώς και μας οδηγούν στο να σκεφτούμε την μεταφορά κονδυλίων και από τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και από άλλες πηγές έτσι ώστε να προστατευτούν ε, αυτά τα κεφάλαια και να διασφαλιστεί η επάρκειά τους. Όσον αφορά βεβαίως ε, την προσέλκυση επιπλέον ε, χρηματοδότησης κεφαλαίων, ιδιαίτερα για εταιρείες ε, που προωθούν την καινοτομία, θα πρέπει να δούμε πάλι αυτό το όριο 100.000 ευρώ και να διασφαλίσουμε ότι δεν ξεχνά μια ολόκληρη συζήτηση όσον αφορά την ε, συνεισφορά των ιδιωτών επενδυτών. Πρόκειται κυρίως για θεσμικούς επενδυτές. Αν βάλουμε πολύ χαμηλά το όριο, καταλαβαίνετε ότι θα μπούμε σε μια συζήτηση με τους ε, επενδυτές, ε, τους ιδιώτες. Και βεβαίως πέρα από ένα ανώταρο ποσό το οποίο θα θέσουμε και εκεί θα προκύψει θέμα όσον αφορά τις ε, συζητήσεις και εκεί βεβαίως ε, μπλεκόμαστε και με ε, τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τώρα, όσο περισσότερα άτομα εμπλέκονται και όσο περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης έχουμε, τόσο πιο ζωντανός θα είναι αυτός ο τομέας. Η συζήτηση για τον ε, ορισμό των χαρτοφυλακίων, δηλαδή το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση, καθώς και οι προθεσμίες, δύο-πέντε χρόνια. Οι περισσότερες ε, εταιρείες, αν θέλετε, μετά από πέντε χρόνια έχουν περάσει την πρώτη φάση. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό όριο είναι η στιγμή που στρέφονται προς ε, τα κεφάλαια αυτά. Σήμερα βεβαίως έχουμε 27 διαφορετικές ε, κατηγορίες, μάλλον ορισμούς για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκεί είναι πολύ δύσκολο κανείς να ξεκαθαρίσει περί τίνος πρόκειται. Θα πρέπει λοιπόν να αποσαφινιστούν όλοι αυτοί οι ρυθμοί. Σε γενικές γραμμές ε, είμαι βεβαίως ε, θετικά διατεθειμένος προς αυτή την πρόταση. Πιστεύω ότι πρέπει να ανοίξει αυτή η αγορά κεφαλαίων στην Ευρώπη και πολλά άλλα θέματα παραμένουν εκκρεμή όπως παραδείγματο χάρη η μέση απόδοση αυτών των κεφαλαίων. Αυτό ενδιαφέρει τους επενδυτές. Και θα συμφωνήσω εδώ με τον Σαΐντ ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία και τα μέσα που διαθέτουμε στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής και πώς μπορεί κανείς να συμμετάσχει σε μια τέτοια χρηματοδότηση. Ο συνδυασμός όλων αυτών των μέσων, όλων αυτών των εργαλείων, θα πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα περισσότερα κεφάλαια για τις επιχειρήσεις και θα συμφωνήσω εδώ ότι πρόκειται για μια πολύ καλή βάση συζήτησης. Συγχαίρω τους συζητητές και θεωρώ ότι πρέπει ακόμα πολλά να κάνουμε για να δώσουμε περισσότερη κινητικότητα και να προωθήσουμε αυτή την αγορά στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, όπως και με τον προηγούμενο φάκελο. Χαίρομαι για αυτή τη συνεργατική προσέγγιση που έχουμε υιοθετήσει. Γνωρίζω ότι ο εισηγητής είναι πολύ ανοιχτός σε συζητήσεις και σε προτάσεις. Επίσης επικροτώ το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η πρόταση. Είχα ακούσει τις προειδοποίησεις από τη βιομηχανία επιχειρηματικού κεφαλαίου ότι δεν πρέπει να αναμειγνέται με τα hedge funds και όλα αυτά. Για να είμαι δίκαιος προς την Κομισιόν έχει μάθει το μαθημά της και έκανε αυτή την πρόταση. Χαίρομαι λοιπόν γι' αυτό. Πρέπει επίσης να καταλάβουμε το περιβάλλον που υπάρχει εκεί έξω ε, καθώς οι τράπεζες υφίστανται πιέσεις, ε, η δανειοδοτική τους ικανότητα είναι περιορισμένη. Ε, οι εταιρείε τώρα ψάχνουν αναλλακτικέ πηγές και πιστεύω ότι τα επιχειρηματικά κεφάλαια θα παίξουν κάποιο ρόλο σε αυτό. Όσοι απευθύνονται σε εταιρείε επιχειρηματικού κεφαλαίου πρέπει να είναι ρεαλιστικοί στις προσδοκίες τους, Πρέπει να, να καταλάβουν ότι οι επενδυτές συχνά θέλουν απόδοση. Ε, πρέπει να είναι ρεαλιστικές όσον αφορά την προσφορά που κάνουν σε πιθανούς επενδυτές. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η πρόταση θα λύσει τα πολιτισμικά προβλήματα που έχουμε σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, σημαντικό, πιστεύω, ωστόσο βήμα θα αποτελέσει όλο αυτό. Μερικά σημεία που θέλω να αναφέρω. Το πρώτο, όπως ανέφερε ο Φίλιπ, το κατόφλιο των 500 εκατομμυρίων ευρώ και το σήμα ΕΦΚΑ και το MFT και πώς θα συντεριάξουμε όλα αυτά και οι προτάσεις καλό θα ήταν το Ταμείο να επιλέξει κατά πόσο τα θέλει όλα αυτά Ποια είναι η πρότασή σας για να αποφύγουμε οποιασδήποτε αμφιβολίες εγώ δεν είμαι Βέλγος. Ήθελα να το διασαφηνίσω σε περίπτωση που κάποιο δεν το γνώριζε. Χαίρομαι ωστόσο που ο εισηγητή ε, είναι διατεθειμένος να ακούσει κάποιες από τις παρατηρήσεις μου. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Επίσης αυτό το ζήτημα των επενδυτών και ποιου επενδυτέ πρέπει να επιτρέπουμε. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να επιτρέπεται να επενδύουν ό,τι θέλουν όπου θέλουν εφόσον κατανοούν τους κινδύνους. Αυτό είναι όμως το πρόβλημα υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος σε θέματα καταναλωτών. Εάν έρθει κάποιος ψηφοφόρος και μας πει εγώ επένδυσα αυτά, ναι τα διάβασα όλα, τα έγραφα, τα υπέγραψα, αλλά δεν γνώριζα ότι έκανα επένδυση σε κάτι τέτοιο και δεν θέλω να χάσω τα λεφτά μου. Εμείς οι πολιτικοί υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, συνεπώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το ποιον επιτρέπουμε να επενδύσει. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια ευθυγράμμιση με άλλους κανονισμούς και οδηγίες η ιδέα του επενδυτή που πληρεί τις προϋποθέσεις ίσως και η ευθυγράμμιση με άλλες οδηγίες και κανονισμούς και επίσης οποιοδήποτε περιθώριο που μπορεί να παρέχουμε η ευελιξία στις εθνικές αρμόδιες αρχές. Το τελευταίο που θέλω να πω, το τελευταίο ζήτημα είναι το ζήτημα των πέντε ετών. Σίγουρα δεν θέλουμε να βοηθήσουμε μόνο νεοσύστατες επιχειρήσεις αλλά και επιχειρήσεις σε φάση ανάπτυξης Ορισμένες φορές ε, νεοσύστατες επιχειρήσεις έχουν χρηματοδότηση, έχουν σχέδια, αλλά τη στιγμή που μπαίνουν σε φάση ανάπτυξης χρειάζονται χρήματα. Θα ήθελα λοιπόν ο συγητής πολύ προσεκτικά να εξετάσει αυτό τον περιορισμό. Κατά πόσο θέλει να περιορίσει το πεδίο εφαρμογή σε εταιρείε ε, ηλικίε έω 5 ετών. Το άλλο ζήτημα είναι οι θεματοφύλακε. Δεδομένου ότι τα ταμεία αυτά δεν διαθέτουν ε, χρηματοοικονομικά μέσα, συχνά οι απαιτήσει οικονομικού ελέγχου καλύπτουν την προστασία των επενδυτών. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να... για, να είναι απαραίτητο ένα θεματοφύλακα, ε, εκτό αν υπάρχουν άλλε περιστάσει. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Αν κατάλαβα καλά, επειδή μας περασεύει λίγος χρόνος, μπορούμε να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Επικεφαλής δεν είναι Βέλγος. Τίλμαν, έχετε το λόγο. thanks uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μας δίνετε το λόγο. πάρα πολύ θετικές αντιδράσεις. Αυτό μας ε, χαροποιεί γιατί δεν είναι, συμβαίνει πάντα. Και πρόκειται για ένα θέμα το οποίο το συζητούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χαιρόμαστε που φτάσαμε σε μια θετική ατμόσφαιρα συζήτησης. Το θέμα αυτό βεβαίως προκαλεί και κάποιες ανησυχίες. Καταρχήν, όσον αφορά την ελκυστικότητα αυτού του σχήματος, θα πρέπει να είναι ε, λίγο διαφορετική η προσέγγιση μας από αυτή της ε, πρώτης κατηγορίας ε, κεφαλαίων, καθότι δεν θα είναι τόσο θετική αξιολόγηση. Εάν δεν υπάρχει ένα από φορολογικής απόψεως ουδέτερο σχήμα, δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει. Δεν πρόκειται να είναι επιτυχή οι προτάσεις μας. Γι' αυτό και ε, ξέρουμε ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα, αν θέλετε, για να δημιουργηθεί ένα κλίμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή επιχειρηματικού κεφαλαίου ελκυστικού, χωρίς κίνητρα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία να είναι επιτυχής. Όπως σας είπα από την αρχή, θα πρέπει να προτείνουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με το AIMFMD, τους κανόνες αυτούς. Θέλουμε να, να εμβαθύνουμε συγγνώμη, την βάση και αυτό το λεγόμενο διαβατήριο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην είναι περίπλοκο, να μην είναι επαχθές, οι κανόνες να μην είναι δύσκολοι να κατανοηθούν και να εφαρμοστούν και γι' αυτό και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει με έναν δυναμικό τρόπο προτείνοντας αρκετά κίνητρα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιβραδύνουμε το ξεκίνημα αυτού του σχήματος. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό να δούμε κατά πόσο αυτό είναι ελκυστικό ή αποτρεπτικό. Θα ήθελα, όσον αφορά τις τροπολογίες, να πω δύο-τρία πράγματα. Έχουμε βεβαίως διαφορετικούς ορισμούς. Φυσικά η διαφορά μεταξύ των ε, ορισμών εξαρτάται και από το περιεχόμενο, δηλαδή εάν κάποιος επιλέξει ένα συγκεκριμένο ε, τύπο επιχειρηματικού κεφαλαίου, και κατά πόσο μπορεί κάποιος ε, να αποσύρει τα χρήματα που έχει επενδύσει στο τέλος ε, της ε, διαδικασίας, όταν ολοκληρωθεί δηλαδή η επένδυση. Ε, σε καμία περίπτωση βεβαίως αυτά τα ποσά δεν θα πρέπει να παραμείνουν σταθερά και εννοείται ότι παραδείγματο χάνει τα 100.000 ευρώ είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα αυξηθεί. Μιλάμε για τις επενδύσεις, ανοιχτές επενδύσεις, κλειστές επενδύσεις, όταν δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα να αποσύρει κάποιος ε, το κεφάλαιό του ε, στο τέλος της διαδικασίας είτε κατά τη διάρκεια κάποιων άλλων φάσεων. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι σας ανησυχεί επίσης και το θέμα της έδρας αυτών των ε, ταμείων. Η έδρα του διαχειριστή. Διότι αυτός είναι, αν θέλετε, ο εγγυητής των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου. Η επιχείρηση, βεβαίως, υπόκειται κάθε φορά στην νομοθεσία του κράτους. Ο διαχειριστής θα πρέπει εδώ να παρέχει τις συγκεκριμένες εγγυήσεις όσον αφορά τις επενδύσεις το 70% εκεί έχουμε καταλήξει του κεφαλαίου και αυτό βεβαίως είναι μια επιλογή του διαχειριστή. Οι εταιρείε θα πρέπει να βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε δει και όταν λέτε ότι οι προσπάθειές μας είναι να δημιουργήσουμε ανάπτυξη στην Ευρώπη, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και στις περισσότερες περιπτώσεις ή σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει οι έδρες των εταιριών αυτών να βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν ε, συγχωνεύσεις ή συνεργασία με επιχειρήσεις ε, αλλού στον κόσμο. Η συνεργασια με επιχειρησεις όμως όπου δεν υπάρχει κάποια επιχείρηση σε ευρωπαϊκή επικράτεια, σε μία από τις ευρωπαϊκές χώρες, θα πρέπει να αποκλειστεί. Μία θηγατρική θα πρέπει να υπάρχει ή ένα, μια βιομηχανική μονάδα, μια μονάδα παραγωγής η οποία θα πρέπει να βρίσκεται στην Ευρώπη. Αυτά όσον αφορά την έδρα. Τι άλλο, ήθελα να αναφέρω και κάτι άλλο, αλλά το ξέχασα. Προφανώς δεν θα ήταν σημαντικό. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι εξετάζουμε, α ναι, τις σχέσεις το AFMD. Το χαρτοφυλάκιο ενός ε, φορέα που ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια. Στην ε, Ευρώπη, όπως ξέρετε, τα ποσά αυτά φτάνουν μέχρι 60 εκατομμύρια ευρώ. Το σήμα λοιπόν, το ευρωπαϊκό σήμα, τι θα πρέπει να γίνει εάν αυτό το ποσό ξεπεράσει αυτά τα ανώτατα όρια. Αυτό βεβαίως είναι θέμα πολιτικό. Και είτε θα πρέπει να θεωρηθεί μια εξαίρεση, είτε να θεσπιστεί ένας ε, ειδικός κανόνας λέξη specialis για αυτές τις περιπτώσεις. Όταν περνάτε παραδείγματο χάρη το ποσό των 500.000. Τι ακριβώς θα γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Και τελειώνοντας θα ήθελα να σας πω ότι σαφώς και θα πρέπει να αυξήσουμε την ελκυστικότητα του δικού μας συστήματος σε σχέση με το EFMD, ότι θα πρέπει να είναι ένα λεγόμενο light καθεστώς, ότι ο manager, ο διαχειριστής θα πρέπει να προσφέρει κάποιες εγγύησεις και να έχει πλήρη έλεγχο, οι κανόνες για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να παραμείνουν και βεβαίως όλα αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να υιοθετηθούν σε μία ασπεσμένη διαδικασία από το Συμβούλιο και το Σας... Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως θα πρέπει μετά από την Επιτροπή να σας δώσουμε και εσάς το λόγο εάν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι με έχει εντυπωσιάσει πλήρως το επίπεδο λεπτομεριών και γνώσεων για το τι διαμείβεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις εταιρείε επιχειρηματικού επίπεδο. Δεν περίμενα είναι τόσο υψηλό επίπεδο συζήτηση. Θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, τέθηκε λόγος για τις μη εισηγμένες εταιρείε. Όντως, οι εταιρείε που είναι ε, εισηγμένε σε κάποια χρηματιστήρια είναι πολλές χειρότερες από κάποιες μη εισηγμένε. Διότι έχει κανείς την ε, αξιολόγηση ε, των αποθεμάτων, αλλά δεν έχει απαραίτητο ούτε ρευστότητα, ούτε πρόσβαση σε νέα κεφάλαια. Και πολλές τέτοιου είδου επιχειρήσεις δεν μπορούν να επενδύσουν τις συγκεκριμένε εταιρείε. Και πρέπει να πω ότι υπάρχει εξαίρεση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων που μπορεί να παρέχει ε, στις μη βοήθειες της εταιρείε που είναι ρυθμισμένε σε εναλλακτικά χρηματιστήρια, μη καθορισμένα. Μη ρυθμισμένα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο. Πολλέ συζητήσει επίσης αφορούσαν αυτό το κατόφλι των 100.000 ευρώ. Εμείς στι εταιρείε μας, στα pre fund που έχουμε, επίσης επιβάλλουμε το κατόφλι των 100.000. Για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, όπως είπε, και κάποιος όταν πάει κανείς σε έναν ιδιώτη επενδυτή, οι συζητήσεις που κάνει διαφορετικό επίπεδο. Δεύτερον, πρέπει κάποιος να ε, χειριστεί πληροφορίες, να απαντήσει και να έρθει σε συναλλαγές και σε επαφή με 5-10 επενδυτές. Δεν είναι το ίδιο με το 50 ή με 2.500. Και όποιος ιδιώτης θέλει να συμμετάσχει σε τέτοιες εταιρείε μπορεί να αγοράσει μετοχές στην αγορά και αν δεν του αρέσει η επίδοσή μας ή ό,τι κάνουμε μπορεί να τις, ε, πολύ να τις ανταλλάξει και να φύγει. Αυτό λοιπόν είναι καλό. Και αν κατεβείτε κάτω από το κατόφλι των 50-100 χιλιάδων, δεν ξέρω ποιο είναι, είσαστε κάτω από... Υπάγεστε σε άλλου είδους ε, ε, νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν να κάνετε εσείς την περιοχή. Στη, στο Βέλγιο η φλαμανδική κυβέρνηση έδωσε κάποια φορολογικά κίνητρα για την εταιρεία Αρχιμίδης. Ε, υπήρξαν πάρα πολλοί επενδυτές, αλλά σήμερα πολλοί θέλουν να αποσυρθούν από αυτό το επενδυτικό σχήμα γιατί θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα λεφτά τους για κάτι άλλο, γράψουν ένα σπίτι κάτι άλλο. Και αυτό έγινε διότι κατέβηκε το κατόφλι. Τα feeder funds λοιπόν καλά θα προβλέπονται όσον αφορά το κατόφλι των αυτό προβλέπεται για τα πέντε χρόνια θα σας πω ότι βρήκαμε για επενδύσει σε υβριδικά αυτοκίνητα ότι υπήρχε για 20 χρόνια μία βελγική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται ε, εδώ και 20 χρόνια στον τομέα αυτό και μετά τις ε, επενδύσεις που έγιναν χρεοκόπησε διότι υπήρχε κακή διαχείριση. Έτσι στραφήκαμε στην ε, ε, σε μια κινέζικη επιχείρηση και αυξήθηκε κατά πολύ η παραγωγή και άρχισαν οι ε, υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα σιγά σιγά να παράγονται και θα μπουν σιγά σιγά στην αγορά. Πρέπει λοιπόν να είναι καλής πολύ προσεκτικός να κάνει κάτι καινούριο στην αγορά. Ήθελα επίσης να επισημάνω ότι είναι περιττός ο φόρτος όπως επισημάνθηκε. Μιλάμε για capital entrances σε μερίδια δηλαδή του 5% επενδύουμε σε επιχειρήσεις και όλες οι συμμετοχές αυτές είναι καταχωρημένες. Έχουμε έναν οικονομικό ελεγκτή που ελέγχει στα μητρώα της εταιριών κάθε χρόνο κατά πόσο οι μετοχές που έχουμε στα βιβλία μας υπάρχουν όντω και έχουν καταχωρηθεί στα μητρεώτα των εταιριών. Θεωρώ λοιπόν ότι ένας θεματοφύλακας θα είχε περιορισμένη αξία και θα αύξανε υπερβολικά το διοικητικό άχθος. Πολλά συζητήθηκαν σε σχέση με το σύνδεσμο με την οδηγία Alternative Alternative Fund Investment Management. Πιστεύω ότι αυτή η οδηγία έχει κάνει δύο πράγματα στην Ευρώπη. Το ένα που έκανε δημιούργησε μία ε, ε, κοινωνία δύο ταχυτήτων. Στο επιχειρηματικά κεφάλαια κάτω από δύο εκατομμύρια μπορεί κανείς να επιλέξει να βγει, αλλά κατά την άποψή μου Αυτός ο κανονισμός είναι, είναι ήδη πολύ δύσκολο να πείσει κάποιος είναι διευθυντή ενός συνταξιδοτικού τιμίου να, να επενδύσει σε επιχειρηματικά κεφάλαια επειδή είναι επικίνδυνο. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Ωστόσο πρέπει να τους πείσουμε. σε αυτή την κατηγορία των εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων Όλα αυτά τα στοιχεία ρυθμίζονται υπό αυτή την οδηγία. Και ε, σε αυτό το πλαίσιο παρέχουμε επίσης μία επιλογή opt-out. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται ούτε να λάβετε χρήματα, ούτε καν να μπορέσετε να κανονίσετε μια συνάντηση. Εμείς, παρότι γνωρίζαμε αυτό το κατόφλαιο των 500 εκατομμυρίων, αποφασίσαμε να συμμετέχουμε, διότι διαφορετικά θα διακοπεί η παροχή κονδυλίων. Κατά την άποψή μου λοιπόν δημιουργήθηκαν πολίτες δύο ταχυτήτων στην Ευρώπη, αυτοί που συμμορφώνονται με την οδηγία αυτή, το Alternative Fund Management Directive και όσους δεν συμμορφώνονται. Για αυτούς που δεν συμμορφώνονται αυτό το καθεστώς είναι ενδιαφέρον, μπορεί να τους βοηθήσει στην άντληση κεφαλαίων. Αυτό που με ανησυχεί και ίσως θα έπρεπε να το πω στα φλαμανδικά όταν αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει κάποια σύνδεση με τα δημόσια επενδυτικά ταμεία η ύπαρξη ενός διαβατηρίου ή ρύθμισης ε, ως ευρωπαϊκού επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν πρέπει να αποτελεί απέτηση για να λάβει κάποιος χρήματα από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο. Πιστεύω η Κομισιόν σωστά ανησυχεί για το πόσο δημοφιλή θα γίνουν αυτά όταν ξεκινάει κανείς ένα κανονισμό και τη συμμόρφωση όλες οι διευθυντικές ομάδες θα συζητήσουν κατά πώς θα επιλέξουν εναλλακτικά επενδυτικά σχέδια ή κατά πώς θα προτιμήσει περιορισμένη συμμόρφωση υπό αυτό το καθεστώς. Πιστεύω ότι η εμβάθυνση των κεφαλαίων τη ικανότητα μικρών ε, ταμείων επιχειρηματικού κεφαλαίου να αντλήσουν κεφάλαια θα απομένει να αποδειχθεί. Όπως επεσήμανε η Σοφή είναι πολύ ωραία ετικέτα για μάρκετινγκ το να έχει κάποιος αυτό το καθεστώς αλλά δεν θα οδηγήσει απαραίτητα σε μεγαλύτερη ροή κεφαλαίων. Τι άλλο ήθελα να πω. Open-ended και closed-ended, ε, ανοιχτού τύπου και κλειστού τύπου συζητήθηκε. Πολύ καλά επεσήμανε η Κομισιόν όταν χαμηλώνει κανείς το κατόφλιο πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο χρήση ε, μετοχών που είναι εισηγμένε στο χρηματιστήριο. Το Horizon 2020 πολλά χρήματα υπάρχουν και γι' αυτό για την υποστήριξη των καινοτόμων βιομηχανιών μας και εγώ εναπλάκνω σε πολλές συζητήσεις για το μέλλον. Το μόνο που μπορώ να πω εδώ είναι ότι το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο επένδυσε στο Ταμείο μας μέσω του προγράμματος SIP και αυτό βοήθησε εξαιρετικά. 70 ή 80 εκατομμύρια αντλήθηκαν, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο δέσμευσε 50 εκατομμύρια ε, χάρη στην αξιοπιστία του απέκτησε πάνω από 100 εκατομμύρια για ε, καθαρές τεχνολογίες και έτσι είμαστε τους μεγαλύτερους επενδυτές σε αυτόν τον τομέα. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε μία ροή πραγματικά πανευρωπαϊκού επίπεδου. Η συμβουλή μου λοιπόν είναι ότι όταν υπάρχουν πολλά χρήματα που επενδύονται σε ένα πρόγραμμα, πολλοί οργανισμοί, πολλές ομάδες θα θελήσουν να πάρουν μερίδιο της τούρτας. Θα συμβούλευα την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να φροντίσουν να ε, συγκεντρώσουν τα χρήματα και να οικοδομήσουν βάση του πολύ καλού έργου που έχει γίνει από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο στο παρελθόν και όχι να κατακαιρματίσουν υπερβολικά αυτούς τους πόρους. Διαφορετικά δεν θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Νομίζω ότι κάλυψα τις περισσότερες από τις ερωτήσεις που ακούστηκαν. Κατά κάποιο τρόπο, λέει η Πρόεδρος, ο χρόνος έχει αρχίσει και μας πιέζει. Αν έχετε ακόμα ένα ή δύο σημεία. Ναι, εγώ θα είμαι πολύ πολύ σύντομη. Συμφωνώ με τα περισσότερα σχόλια που άκουσα, εκτός ίσως από τα 100.000 το όριο, το οποίο για μένα είναι υψηλό. Δεν πρέπει να μπούμε σε επενδύσεις ιδιωτών. Από τη μία λοιπόν έχουμε αυτό το 100.000 το όριο, από την άλλη βεβαίως για κάποιες μικρές επιχειρήσεις αυτό το 100.000 ίσως είναι πολύ ψηλό ποσό. Τώρα, αυτό το 70% όσον αφορά το όριο για τις επενδύσεις, αυτό εξαρτάται για το πώς το μετράμε και πώς το καθορίζουμε. 70% πλήρης επένδυση στην αρχή του ταμείου, όταν ολοκληρωθεί η επένδυση στο ταμείο. Αυτό εξαρτάται και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αυτό το ποσοστό 70% να αντιμετωπίζεται στο τέλος κάθε χρόνου. Ένα άλλο θέμα είναι η έδρα των ε, εταιριών χαρτοφυλακίου. Αυτό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιοριστεί σε εταιρείες ευρωπαϊκές, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πλειοψηφία των επενδύσεων σαφώς και θα πρέπει να απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι κάποιες άμεσες επενδύσεις αλλού στον κόσμο δεν μπορεί να έχουν θετικές επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε λοιπόν να το αποκλείσουμε 100% ότι κάποιες από αυτές τις επενδύσεις θα γίνονται και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Φιλίπ. Θα είμαι σύντομος. Πολύ χρήσιμε όλε οι πληροφορίε που μα έδωσαν οι ομιλητέ μα. Ε, σίγουρα θα τι λάβουμε υπόψη. Λοιπόν, υπάρχει αρκετά ευρεία συνένεση εδώ και θα προσπαθήσω να εργαστώ προ αυτή την κατεύθυνση Όσον αφορά τον κανόνα των 5 ετών, προφανώ δεν είναι σωστό κανόνα για να επιτύχουμε το στόχο. Στόχο είναι να πάνε αυτά τα κονδύλια σε νέα εγχειρήματα, σε νέα επιχειρηματικά κεφάλαια, όχι σε παραδοσιακέ εταιρείε. Είτε μιλάμε για εταιρείε εδώ που πραγματικά επιχειρούν κάτι καινούριο ή νέε εταιρείε. Η ερώτηση που θα σας κάνω ανεπίσημα είναι πώς θα είμαστε βέβαιοι ότι θα παραμείνουμε στον τομέα των επιχειρηματικών κεφαλαίων, ε, κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. Πολλά άλλα σχολεία που άκουσα θα τα λάβω υπόψη. Το θέμα όσον αφορά το θεματοφύλακα δεν είμαι μετακίνητο σε αυτή την ιδέα. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς ε, γίνεται εδώ πέρα. Θα ήθελα να δω τις τροπολογίες σας και πιστεύω θα είναι εύκολο να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό. Πιστεύω λοιπόν ότι όλη η διαδικασία θα είναι αρκετά ομαλή. Πολύ καλά, σας ευχαριστούμε. Θα θέλω να ευχαριστήσω τους προκεκλημένους μας. Λοιπόν, προθεσμία κατάθεσης 20 Μαρτίου παρολίες, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 28 το μεσημέρι. Εξέταση των τροπολογιών 24-26 Απριλίου με προβλεπόμενη ψηφοφορία στην Επιτροπή τέλος Μαΐου, 30-31 Μαΐου και ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Πρόκειται για μια ταχεία διαδικασία. Ευχαριστώ. Έχουμε κερδίσει σχεδόν πέντε χρόνια. Συγγνώμη, πέντε λεπτά. Uh, από το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Λοιπόν, περιμένουμε να φύγουν κάποιοι από την αίθουσα. Υπότιτλοι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 Okay, if we could... Λοιπόν, παρακαλώ να ξαναρχίσουμε. Φιλίπ! Συνεχίζουμε με το show του Φιλίπ Λαμπέρ. Σημείο 8. Οι Ευρωπαϊκές Ενεργειακές Υποδομές και κατάργηση της απόφασης 1364 Παύλα 2006 Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Γνωρίζετε όλοι, σίγουρα περί τίνος πρόκειται. Επί της ουσίας είναι υπεύθυνη ήτρε. Η Άννη είναι, αν θέλετε, συγγήτρια επί της ουσίας στην Επιτροπή Ήτρε. Εγώ πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Δεύτερη εισήγηση την ίδια μέρα. Ευχαριστώ πολύ και πραγματικά πρόκειται για κάποια από τα τμήματα του θέματος αυτό που πρέπει εμείς να επεξεργαστούμε. Δεν θέλω να μπω στην λεπτομέρεια. Χρηματοδότηση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, τις υποδομές, δίκτυα μεταφοράς και πρόκειται για την επιλογή των προτεραιοτήτων, κριτήρια επιλεξιμότητας. Έχω δύο τροπολογίες, μόνο δύο τροπολογίες. Πρώτον, όσον αφορά, αν θέλετε, την επιλογή των προγραμμάτων, πάντα να έχουμε κατά νου την Ευρώπη 2020. Ίσως έχω ε, πολλές φορές αναφέρει το θέμα αυτό, αλλά πραγματικά δεν πρέπει να ξεχάσουμε σε καμία νομοθετική πρόταση τους στόχους αυτούς. Γι' αυτό και πρέπει να συνδεθεί το θέμα αυτό με τους στόχους ε, του 2020. Επίσης, ένας από τους πολύ σημαντικούς στόχους αναφέρεται στην ενέργεια. Δίκτυα ενέργειας που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ξέρετε ότι η Γερμανία επέλεξε να αποδεσμευθεί από τον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Αυτό έχει πολύ συγκεκριμένες επιπτώσεις και βεβαίως συγκεκριμένα για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα πρέπει λοιπόν να προετοιμάσουμε όλες αυτές τις αποφάσεις, ιδιαίτερα να εξεταστούν οι επιπτώσεις Κάναμε μία τροπολογία και βεβαίως έχουμε μία συζήτηση που έχει ξεκινήσει με την ε, Επιτροπή. Δεν τους βλέπω όμως εδώ. Κάπου θα είναι οι εκπρόσωποι της Επιτροπής. Δεν ξέρω, ίσως η συζήτηση δεν έχει ολοκληρωθεί, θέλει ακόμα επεξεργασία το θέμα αυτό. Είχα μια πολύ έντονη συζήτηση ακριβώς πριν ξεκινήσει αυτή η συνάντηση όσον αφορά την αύξηση του κόστους ενός προγράμματος το οποίο αν ξεπεράσει το 30% μάλλον αν η αύξηση του ποσού ξεπεράσει το 30% θα πρέπει να επανεξεταστούν όλα τα κριτήρια της επιλεξιμότητας. Ε, το θέμα είναι ότι ουσιαστικά αν κάτι τέτοιο συμβεί πρόκειται απλά για κακό σχεδιασμό. Ο κακός σχεδιασμός λοιπόν δεν μπορεί να θεωρηθεί κάτι το συνηθισμένο και κάτι το οποίο θα το θεωρήσουμε σαν business as usual. Αυτός λοιπόν ο κανόνας, ο οποίος ουσιαστικά ενσωματώνεται στην νομοθεσία, δεν είναι κάτι το αυστηρό, ίσως κάποιοι το χαρακτηρίζουν αυστηρό, αλλά η αύξηση του ποσού κατά 30% δεν μπορεί να θεωρηθεί κάτι το κοινό ή το ε, συνηθισμένο. Χρειάζεται κάποια πειθαρχία. Προσπαθούμε να επιβάλλουμε πειθαρχία στα κράτη. Ας, ας επιβάλλουμε πειθαρχία και στον ιδιωτικό τομέα και στις αγορές. Η πρόταση αυτή αναφέρεται σε υποδομές, υποδομές κάθε είδους ενέργειας. Εδώ θα πρέπει ιδιαίτερη σημασία να δοθεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν είμαι βέβαιος ειδικό, αλλά αν υπάρχουν κάποιοι που είναι εμπειρογνώμονες, θα ήμουν βεβαίως πολύ ευτυχής να συνεργαστώ. Θα σε ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ε, ναι, πρόκειται εδώ για μια πρόταση που αφορά τις εξελίξεις ε, ουσιαστικά στους ε, τομείς ε, της ενέργειας, τα δίκτυα και τις υποδομές. 200 εκατομμύρια ευρώ είναι οι ανάγκες επενδύσεων για τις υποδομές για τα επόμενα 8 χρόνια. Και βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι οι υποδομές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφορά σε τομείς όπως ε, το φυσικό αέριο, 70 εκατομμύρια στον τομέα αυτό και βεβαίως το θέμα της αποθήκευσης η επί της Επιτροπή είναι η Επιτροπή Ήτρε. Έχουμε μελετήσει τις ε, προτάσεις και βεβαίως αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος Λάμπερτς είναι καθαρά θέματα χρηματοδότησης, πάρα πολύ σημαντικά. Οι υποδομές μεταφοράς ενέργειας. Βλέπουμε εδώ συγκεκριμένες ε, ελλείψεις. Βλέπουμε πρωτοβουλίες, 12 αν θυμάμαι καλά. Το πρώτο βήμα για μένα θα πρέπει να είναι αν αυτοί οι διάδρομοι που έχουν επιλεγεί για τη μεταφορά είναι σωστά, σωστές επιλογές. Και κατόπιν οι 12 προτάσεις για αυτές τις ε, υποδομές, ιδιαίτερα με ενδιαφέρει και το θέμα του διοξιδίου του άνθρακα νέες τεχνολογίες στον τομέα του άνθρακα και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι εδώ οι πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Τα δίκτυα διοξιδίου του άνθρακα, όπως ξέρετε, εδώ πρόκειται για κάτι το οποίο αφορά ιδιαίτερα τις βόρειες χώρες, μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Νορβηγίας, παραδείγματος χάρη, και βάσει των στοιχείων που έχουμε από την αντίστοιχη εταιρεία της Νορβηγίας. Εδώ πρόκειται για πολύ συγκεκριμένες μεταφορές από την Μεγάλη Βρετανία, την Γερμανία, τις κάτω και κοίταξα πολύ προσεκτικά αυτά που προτείνουν οι Νορβηγοί. Οι Νορβηγοί ουσιαστικά έχουν ένα φυσικό αέριο και αν θέλετε το 9,5 αυτής ε, της ε, αυτών των εκπομπών χρησιμοποιείται και αν αναπτυχθούν όπως ε, προβλέπεται να γίνει οι νέες αυτές τεχνολογίες, βλέπουμε ότι οι στόχοι που έχουμε θέσει για το διοξίδιο του άνθρακο θα είναι υλοποιήσιμοι. Και εδώ βεβαίως έχουμε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη ε, προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι το οποίο ιδιαίτερα μας αφορά επίσης είναι τα δίκτυα υψηλής έντασης και η αποθήκευση. Έχουμε βεβαίως εδώ κονδύλια σε περιφερειακό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο και συγκεκριμένα κριτήρια και συντελεστές ε, για την ε, υιοθέτηση αυτών των μέτρων. Δεν θέλω τώρα βεβαίως να μπω σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, δεν είμαστε η αρμόδια επιτροπή, αλλά βλέπω αυτό τον κατάλογο κριτηρίων και θα ήθελα να σας πω ότι εκεί βρίσκεται η ουσία. Η παλιά οδηγία έχει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και θυμάμαι τη συζήτηση που είχε γίνει τότε. Υπήρχε η ομάδα Κάρεν Βαν Μίρτ που είχε, αν θέλετε, την αρμοδιότητα, ήταν ο επίτροπος ε, αρμόδιος για θέματα ανταγωνισμού. Πολύ συγκεκριμένες προτάσεις είχαν ακουστεί τότε, γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να προτείνω να συνεργαστούν οι δύο επιτροπές, καθότι πραγματικά χρειάζεται να υπάρξει ομοφωνία, τουλάχιστον να μην υπάρξουν αντικρουόμενες προτάσεις. Βεβαίως οι στόχοι 2020 είναι πολύ σημαντικοί, αλλά κυρίως χρειαζόμαστε μία σταθερή υποδομή η οποία θα ανταποκρίνεται στον σχεδιασμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βεβαίως ότι ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα. Υπάρχουν λοιπόν πολύ σημαντικές προτάσεις, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιες λήψεις που θα έπρεπε να επεξεργαστούμε. Σας παρακαλώ, η προθεσμία για τις τροπολογίες να μην είναι πολύ νωρίς για να προλάβουμε πραγματικά να επεξεργαστούμε το κείμενο, το κείμενο και να κάνουμε επικοδομητικές προτάσεις. Ίσως λοιπόν μετά τις διακοπές του Πάσχα. Ευχαριστώ. 28 Μαρτίου λέει εδώ μπροστά μου η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Θα ζητήσουμε λοιπόν από τη Γραμματεία κάτι να κάνει εδώ. Άννη. Ευχαριστώ πολύ Σάρον και ευχαριστώ πολύ και τον ε, εισηγητή μας, τον Φιλίπ ε, Λάμπερς. Δυστυχώς, Φιλίπ, ε, δεν είμαι εισηγήτρια στο πλαίσιο της Επιτροπής Ήτρε, γιατί είμαι πρώην μέλος της Επιτροπής Ήτρε, δυστυχώς. Χαίρομαι που βρίσκομαι μεταξύ συναδέλφων καλών από την Επιτροπή Ήτρε, αλλά εγώ έπρεπε να παρετηθώ στο πλαίσιο εσωτερικών αλλαγών της αντιπροσωπείας μας. Παρ' όλα αυτά ε, είμαι η σκιώδης ε, εισηγήτρια στην ε, γνωμοδότηση του, του Φίλιπ και θέλω με την ευκαιρία να τον συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά του. θεωρώ ότι η συντριπτική πλειονότητα των τροπολογιών που έχει επεξεργαστεί και έχει υποβάλει είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αξίζει να υποστηριχθούν και θα αναφέρω ειδικότερα αυτές που προάγουν τα περιβαλλοντικά ωφέλη και εστιάζουν στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση σε 20%. Είναι οι τροπολογίες 4, 21 και 22. Οι τροπολογίες που συμβάλλουν στην κατάρτιση και στην συμπερίληψη των εφιών δικτύων στα χρηματοδοτούμενα έργα οι τροπολογίες 20 και 26 ε, και βεβαίως οι τροπολογίες είναι μια ε, πολύ σωστή πρόταση ε, αυτή που αφορά την ανάγκη επιμερισμού των κερδών από την λειτουργία των έργων υποδομών σε αναλογία με τον επιμερισμό του κόστους κατασκευής τους μεταξύ των φορέων υλοποίησης. Ε, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας το επεσήμαναν και οι προλαλήσαντες το ευρωπαϊκό δίκτυο βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, ε, προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το στόχο ε, του 2020 σε ό,τι αφορά το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση αλλά και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι σαφές ότι εάν δεν γίνουν έργα υποδομών για την αποτελεσματική σύνδεση περιοχών που παρουσιάζουν ένα πλούσιο, εξαιρετικά πλούσιο δυναμικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έργα λοιπόν υποδομής εκεί και διασύνδεσης με το ευρωπαϊκό δίκτυο, ε, πιθανό να θέσουμε σε κίνδυνο ε, την επίτευξη του στόχου αυτού μαζί με τα οικονομικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά ωφέλη που τον συνοδεύουν ο εισηγητής έχει εντοπίσει και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου τη σύνδεση των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας με την στρατηγική ευρώπη 2020 και με τους στόχους για την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας. με δεδομένο ότι κουβεντιάζουμε για την γνωμοδότηση της επιτροπής οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων ε, θα ήθελα ε, σε μία πρόταση να εστιάσω την προσοχή μου και να ζητήσω τη γνώμη του εισηγητή βεβαίως και των συναδέλφων το γεγονός ότι στις συνθήκες οικονομικής κρίσης που βρισκόμαστε σήμερα υπάρχει έντονη διαφοροποίηση της πιστοληπτικής ικανότητας ανάμεσα στα κράτη μέλη και σε πιθανούς επενδυτές και αυτή η έντονη διαφοροποίηση μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπίες και σε σημαντικά εμπόδια στη χρηματοδότηση των έργων ε, υποδομών με δεδομένο τον ε, ενισχυμένο τον αυξημένο ρόλο που θα έχει ο ιδιωτικός τομέας στη χρηματοδότηση αυτών των έργων. άρα λοιπόν η άρση ε, αυτών των ανισορροπιών θεωρώ ότι είναι κεντρικής ε, σημασίας για να μπορέσουν να προωθηθούν αποτελεσματικά και ισορροπημένα ε, σε όλη την ευρωπαϊκή ένωση οι υποδομές που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων αυτού του κανονισμού. Και μια τελευταία παρατήρηση, το είπε και ο Φίλιπ, αφορά στη διαδικασία επιλογής των έργων στρατηγικής σημασίας των έργων κοινού ε, ενδιαφέροντος θέλω να τονίσω και εγώ από την πλευρά μου ότι η κατανομή της κοινοτική χρηματοδότησης πρέπει να γίνει ε, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται ε, να αποφευθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ έργων που έχουν την προοπτική να συμβάλλουν στην υλοποίηση του ίδιου διαδρόμου προτεραιότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Ε, θα μιλήσω εγώ για το Άλντε. Φίλιππα, νόμιζε ότι δεν γνώριζε τίποτα. Γι' αυτό εγώ μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι γνωρίζω ακόμα λιγότερα. Ωστόσο, πολλά από τα σημεία που ανέφεραν τα μέλη μου φαίνονται αρκετά σημαντικά. Θα μπορέσουμε λοιπόν να τη συζητήσουμε με το Σκιώδη εισηγητή στην ομάδα μου. Θα ήθελα να διερευνήσουμε περισσότερο αυτό που είπες Φιλίπ σε σχέση με το κόστος. Συμφωνώ μαζί σου ότι αν τα πράγματα ξεπεράσουν τον προπολογισμό θα πρέπει να εξεταστούν. Δεν θα έλεγα ότι πρόκειται για αυτόματη περικοπή βέβαια, αλλά σε υποστηρίζω σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό που αναρωτιόμουν είναι ποια ήταν η αλληλεπίδραση μεταξύ πραγματών που γίνονται στο πλαίσιο μειοδοτικού διαγωνισμού που φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία που φοβίζει ορισμένους και διώχνει ορισμένους ε, ε, πιθανούς επενδυτές και κατά πόσο υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ αυτής της διαδικασίας και των περιπτώσεων υπέρβασης του προπολογισμού. Δεν θα ήθελα να Υπάρχει μια τροπολογία. Θα ήθελα μια τροπολογία όπως την προτείνεις ότι αν κάτι αρχίζει να γίνεται διπλάσιο σε κόστος ε, και σε πολυπλοκότητα θα έπρεπε να εμπίπτει στο πλαίσιο μηδιωτικού διαγωνισμού. Ωστόσο, αν είναι πολύπλοκο και ακριβό, μπορεί να μας δίνει καλύτερες απαντήσεις. Εδώ σκέφτομαι δυνατά, μεγαλό, μεγαλόφωνο ουσιαστικά. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία σε αυτό επίσης. Ενημερώνω ότι η γραμματεία μετά από υπολογισμούς λέει ότι θα μπορούσαμε να αναβάλουμε την προθεσμία για τροπολογίες μέχρι την 11η Απριλίου αντί για την 28η Μαρτίου. Θα εξετέσουμε τις ε, τροπολογίες της 30 Μαΐου και μετά θα ψηφίσουμε την 31η Μαΐου που μας δίνει αρκετό χρόνο για την 20η Ιουνίου που θα ψηφιστεί στην ε, αρμόδια επιτροπή. Φιλίπ, έχει το λόγο. Ναι, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Για να είμαι ειλικρινή, κοιτώντα τώρα αυτή την επιτροπή και το φόρτο εργασία τη, αναρωτιέμαι πραγματικά κατά πόσο είναι έξυπνο να ζητήσουμε γνωμοδοτήσει για τόσα άλλα πράγματα. Πιστεύω ότι η συζήτηση, Βέρνερ, για τόσα πολλά σημεία θα μπορούσε να συζητηθεί στην Ήτρα χωρίς πρόβλημα. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να το συζητάμε σε τόσες πολλές ε, επιτροπές, ειδικότερα δεδομένου του φόρτου εργασία της ΕΚΟΝ. Ε, με ανησυχεί βέβαια, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, αλλά αυτή είναι η πρώτη μου αντίδραση. Δεύτερον, όσον αφορά την παρατηρήση τη προθεσμία, δεν έχω πρόβλημα, αλλά Βέρνερ και πάλι εσύ ζήτησες ε, γι' αυτό είναι ότι τα πράγματα δεν προλαβαίνουν να γίνουν, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά όσο παρατείνουμε τα πράγματα ε, για περισσότερο χρόνο, τόσο περισσότερο ε, χώρο χρειαζόμαστε, περιθώριο στη γραμματεία και ούτω καθεξής. Μήπως θα μπορούσαμε να το κάνουμε αμέσως στην Ήτρε αντί για την εικόνα. Ε, αν θέλει να κάνουμε τροπολογίε και οι δυο μα ε, συμμετέχουμε σε αυτέ τι επιτροπέ. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί δεν μπορούμε να εργαστούμε απευθεία στην Ήτρε. Well, we, we, we could put a kind of... Uh, Θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση. Ο Βέρνερ όμως θέλει κάτι να πει. Ίσως ο συνάδελφο, ο Λάμπερτ, έχει μεγάλο φόρτο εργασία σαν έχει πολλέ εκθέσει να κάνει στους πρασίνους. Αλλά αν πιστεύει κανείς ότι είναι άχρηστη η έκον, κάποια θέματα δεν θα τα λάβουμε υπόψη. Εγώ δεν, δεν θα ληφθούν υπόψη. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί του. Ίσως θα πρέπει λίγο να δούμε πώς θα χειριστούμε τις προθεσμίες, αλλά έχουμε και τις διακοπές του Πάσχα. Ας παρατείνουμε την προθεσμία για όπω όπως είπε και η Πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι σε μια επιτροπή είναι σωστό μόνο οι συγητής και οι σκιώδες να παίρνουν το λόγο. Όλος ο κόσμος σε μια επιτροπή, όλοι οι συνάδελφοι είναι σημαντικοί. Άκου, εγώ συμφωνώ όπως είπες όμως, το πραγματικό πρόβλημα είναι τα θέματα αυτά που αφορούν την Ευρώπη να τα εξετάζουμε όλοι. Σωστά. Λοιπόν, Φιλίπ, θα κάνουμε στην συνεδρίαση των συντονιστών. Εμείς συζητούμε άλλα θέματα τα οποία θεωρούμε σημαντικά και αν υπάρχουν κάποια θέματα που πιστεύουν ότι ενδιαφέρον τις πολιτικές ομάδες είναι σημαντικά, τα εξετάζουμε. Πρέπει να πω ότι, όπως σας είπα, 11 Απριλίου η προθεσμία κατάστροπολιών, ώστε τις διακοπές του Πάσχα να τις δουλέψει ο Βέρνερ και εξέταση των τροπολογιών 30 Μαρτίου, ψηφοφορία, Μαΐου, ψηφοφορία 31 Μαΐου. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του θέματος 8 και στα διάφορα ο Ζωαπόλ θέλει κάτι να πει. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Από τις 9 το πρωί, με μεγάλη ευχαρίστηση είμαι στην Επιτροπή θα ευχαριστώ τους διερμηνείς που ήταν το πιο πιστό μας και πολύ άριθμο κοινό από σήμερα το πρωί. Και ακούστε, και εγώ έχω πρόβλημα διερμηνείς. Εδώ έχουμε την ε, ευκαιρία να ακούμε τους διερμηνείς μας, αλλά όταν ε, υπάρχουν ε, τριμερείς και τεχνικές συνεδριάσεις δεν έχουμε διερμηνείς. Για πρώτη φορά χρειάστηκε να ζητήσω, όπως μπορώ να το κάνω, ο συντονιστής έναν διερμηνέα, ο οποίο ψιθυριστά να μου λέει πριν τον αλλά δεν είναι η καλύτερη λύση. Όταν επί ώρες συζητούμε θέματα τα οποία έχουν υποβληθεί στα αγγλικά. Είναι θέμα δημοκρατία στην Ευρώπη. Εκτό να ζητήσουμε σε όλου του ευρωβουλευτέ να περάσουν εξετάσει γλωσσομάθεια σε 14 σε 16 τουλάχιστον γλώσσα, μην πω 23. Είναι λοιπόν απαραίτητο αν θέλουμε να δουλεύουμε ενώ να έχουμε στη διάθεσή μας τους διερμηνείς. Μιλάμε για την Ευρώπη της ποικιλομορφίας και η γλώσσα είναι ένα από τα στοιχεία αυτά. Στα πλαίσια του εξορθολογισμού των δαπανών υπάρχουν κάποια παράλογα πράγματα. Εάν θέλει κάποιος να μειώσει τις δαπάνες, ας μειώσει τα ταξίδια κάποιων συναδέλφων στη Βυρμανία, που δεν ξέρουμε ούτε τι έκαναν, ούτε μας ενημερώνει κανείς, για 3-4 μέρες φεύγουν, παίρνουν και κάποιους διερμηνείς και εμεί τι κάνουμε εδώ. Έχουμε χωρίς καμία βοήθεια εκ μέρους των διερμηνέων 300-400 σελίδες κείμενα να διαβάσουμε. Αν λοιπόν δεν διορθούν τα πράγματα θα σταματήσουμε να δουλεύουμε κι εμείς. Και ο πρόεδρος και το ε, Προεδρείο ας κάνει τη δουλειά που κάνουμε εμείς. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να είμαστε εδώ για ώρε. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά σε αυτήν την Επιτροπή, όπω και σε άλλε. Και είναι απαραίτητη η βοήθεια των διερμηνέων για να φέρουμε σε πέρα στη δουλειά μα. Πιστεύω λοιπόν ότι του χρειαζόμαστε και ελπίζω ότι θα διαβιβάσετε αυτά τα οποία λέγω και στον Πρόεδρο και στο Προεδρία. Ναι, Δεν ξέρω ότι θέλει να μιλήσει ο Βέρνερ. Ναι, θα ήθελα να πω ότι έχει δίκιο ο Ζαν Πολ για δύσκολα θέματα, γνωμοδοτήσεις ε, νομοθετικού περιεχομένου. Χρειαζόμαστε γραπτά κείμενα στην ε, μητρική μας γλώσσα, αλλά και διερμηνία. Θεωρώ πραγματικά ότι για τόσο δύσκολα θέματα, για τόσο αντιφατικά πολλές φορές ε, θέματα και σήμερα που το Κοινοβούλιο έχει πρόεδρο Γερμανό και όταν βλέπω ότι όλα οδεύουν προς ε, μία μόνο γλώσσα, την αγγλική, αυτή της Προέδρου, δεν θέλω να πω τίποτα κακό για αυτή τη γλώσσα, αλλά πραγματικά το πρώτο ταξίδι προς την Βυρμανία, Μπούρμα ή Μιαμάρ, που έλαβε χώρα με τη δική μου Προεδρία, ήταν το πρώτο ταξίδι, η πρώτη επίσκεψη μετά από 50 χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρξαν δύο διερμηνείς, γιατί δύο συνάδελφοι ζήτησαν, δύο γλώσσες έπρεπε να μεταφραστούν. Αν υπήρχε και ένας Γάλλος ε, βουλευτής μαζί μας, θα είχαμε και έναν ε, διερμηνέα σίγουρα για τα γαλλικά. Αλλά δεν νομίζω ότι το παράδειγμα της Βυρμανίας είναι καλό. Υπήρξαν άλλες αντιπροσωπείες με 12 γλώσσες, 12 διερμηνείς, μεγάλα ταξίδια. Για τη Βυρμανία πραγματικά το παράδειγμα δεν ήταν καλό. Κοιτάξτε, δεν ήμουν σαφής. Δεν εννοούσα ότι δεν έπρεπε να πάνε διερμηνείς στη Βυρμανία. Εγώ απλώς αναρωτήθηκα αν έπρεπε ναι ή όχι να γίνει αυτό το ταξίδι. Εκεί ήταν το ερώτημά μου. Μήπως πρέπει να ξαναδούμε λίγο τα ταξίδια και τις επισκέψεις που κάνουμε. Δεν αμφισβήτησα την παρουσία των διερμηνών, ούτε ήξερα πώς ήταν παρόντες. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, Ζαν Πολ. Σε υποστήριξα στο έτοιμά σου για διερμηνία, όπως θα σε έχει ενημερώσει η γραμματεία. Όντως ε, κάνουμε πολλή δουλειά και είναι αρκετά σοβαρά τα πράγματα και χρησιμοποιούμε ελάχιστου διερμηνεί τη δευτερεύουσε εντό εισαγωγικών συνεδρία εργαζόμαστε σε μία είτε σε δύο ή τρει γλώσσε μόνο. Που πιστεύω παρέχει ευνοϊκού όρου για ορισμένου. Ε, Μερικέ φορέ έχουμε αντιπροσωπεία στο Χονγκ Κόνγκ και στη Σιγκαπούρη χωρί κανένα διερμηνέα. Τίνουμε να χρησιμοποιούμε όλο και λιγότερους. Ε, θα είχα πρόβλημα ρατσιστική αντιμετώπιση με τον ε, πρόεδρο όσον αφορά όλο αυτό το ζήτημα της αναδιοργάνωσης και των ταξιδιών με τις αντιπροσωπείες ε, που φαίνεται να επηρεάζει τις εργασίες αυτής της Επιτροπής. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφέρει σε αυτά τα σημεία στη ανοιχτή Επιτροπή ώστε το κοινό να το γνωρίζει αυτό. Άνι, μπορείς να μιλήσεις, ε, αν και θέλω να αφήσω τους διερμηνείς να φύγουν. Όσον αφορά τα όσα είπε ο Ζαμπόλ, συμφωνώ απόλυτα. Απλά ήθελα να σας ε, ενημερώσω ότι γίνεται συζήτηση στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήδη έχει ληφθεί μια απόφαση, όχι να επανεξεταστεί, αλλά να αναζητηθεί να αναζητηθούν ισχυρά θεμέλια όσον αφορά τις αποστολές και τα ταξίδια που πρόκειται να κάνουμε στο εξή ε, σε σχέση με την εξοικονόμηση που πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η Άννη ε, φυσικά είναι αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Να, μια ερώτηση στην Αντιπρόεδρο. Το Προεδρείο που παίρνει αποφάσεις κατά της διερμηνίας έχει ελέγξει εκτός της μετάφρασης και της διερμηνίας πόσες επιπλέον θέσεις έχουν δημιουργηθεί. Πάνω από 500. Πάνω από 500 διοικητικές θέσεις. Αναρωτιέμαι αν όλες αυτές θα καλυφθούν από κάποιον. Ε, δεν γνωρίζω κατά πόσο ο κύριος Λάγκερ μιλάει για νέες θέσεις εργασίας ε, στο πλαίσιο της μετάφρασης, διότι δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο γενικότερα. Το ζήτημα είναι ότι έχει ληφθεί απόφαση εξυγίανσης εξορθολογισμού των δαπανών μας, ανεξαρτήτως ε, του αν αυτές αφορούν μεταφράσεις, αποστολές, ταξιδιωτικές δαπάνες. Ε, είναι μια θέση επί της αρχής υπό τις τρέχουσες προϋποθέσεις μπορούμε να συμφωνήσουμε για αυτή την αρχή και το Προεδρείο είναι ανοιχτό μυαλό, μπορεί να ακούσει τις προτάσεις και τις συστάσεις των μελών. Η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Είμαι βέβαιη ότι ευχαρίστως θα ακούσουμε τα σχόλιά σας και συστάσεις δικές σας. Ευχαριστώ. Ε, ωραία, ευχαριστούμε. Τα υπόλοιπα λοιπόν θα συζητηθούν στο κατάλληλο φόρουμ. Ευχαριστώ τους διερμηνείς. Όπως βλέπετε, νοιαζόμαστε για σας και θέλουμε να σας έχουμε μαζί μας. Ε, θα σας δούμε λοιπόν αύριο το πρωί. Ευχαριστούμε.